Ladies and gentlemen, good Κυρίες και κύριοι καλησπέρα. Καθίστε παρακαλώ γιατί θέλουμε να αρχίσουμε την τακτική μας συνεδρίαση. Η γραμματεία σας μοίρασε ήδη την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρξουν σχόλια θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται η σημερινή ημερήσια διάταξη. Προσθέτω όμως ότι μεταξύ των ομιλητών στον δεύτερο γύρο έχουμε και κάποιον πρόσθετο τον εκπρόσωπο της Ουκρανικής αποστολή στην Ένωση, του πρεσβευτή δηλαδή, που θα μας πληροφορήσει για τα τεκτενόμενα εκεί. Θα ήθελα επίσης να σας πληροφορήσω ότι αν και καταρχάς προσπαθούμε να χορηγούμε διερμηνία για όλες τις γλώσσες των μονίμων και πλήρων μελών της υποεπιτροπής μας που αν δεν απατώμε λέγεται ασφάλεια και άμυνα. Σήμερα έχουμε προβλήματα με τα σουηδικά και το μάθαμε πριν από πολύ λίγη ώρα. Λυπάμαι γιατί δεν θα υπάρξει σουηδική διερμηνία, ούτε κροατική δυστυχώς. λόγω του μεγάλου αριθμού συνεδριάσεων που γίνονται παράλληλα σε αυτό το κτίριο και δεν μπόρεσε η Γενική Διεύθυνση Διερμηνίας να μας χορηγήσει τους πόρους. Την επόμενη φορά όμως θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Σας υπενθυμίζω ότι η συνεδρίαση ως συνήθως αναμεταδίδεται στο web stream. Επίσης πρέπει να λάβατε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης 11, Σεπτεμβρίου αν και για αυτά δεν ακουστεί καμία ένσταση μέχρι να τελειώσει η συνεδρίαση θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Τώρα επιτρέψτε μου να περάσω αμέσως στο πρώτο ουσιώδες σημείο της ημερησίας διάταξης, δηλαδή να καλωσορίσω τους δύο ομιλητές. Αριστερά μου πρώτα είναι ο κύριος Δενιροζέ, που είναι διευθυντής στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας και επικεφαλής μιας καινούργιας διεύθυνσης μέσα στην υπηρεσία αυτή που ασχολείται με την καινοτομία και τη συνεργασία ή συνέργεια. Είναι υπεύθυνο για το κύριο σημερινό μας θέμα η έρευνα σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα. Και ο δεύτερος ομιλητής είναι ο κύριος Βίκτορ Κάρσκι, επικεφαλής της μονάδας στο EEAS, της μονάδας του. Α, όχι, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν, Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και είναι και υπεύθυνο για την άμυνα τέλεια. Θα μας πληροφορήσει για το... θα μας μιλήσει για το δεύτερο θέμα μετά από τον κύριο Ροζέ για την έρευνα λοιπόν σχετικά με την άμυνα και ασφάλεια. Ορίστε κύριε Ροζέ μου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, ε, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Επιτροπή σα και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης είναι πλέον συνήθεια και χαίρομαι διότι θα σας ε, πω για το όραμά μα, για το μέλλον της ε, ε, κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Καταρχά, ε, θα ήθελα να ποτίσω φόρο τιμή ε, στην βοήθεια που έχετε παράσχει στην υπηρεσία το τελευταίο διάστημα. Μα βοήθησε να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό κλίμα και αυτό διαπιστώθηκε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2013. Κάποιοι από εσά κρίνουν τα συμπεράσματα αυτά αρκετά μετρημένα ε, αλλά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου κατάφερε να ε, ξαναβάλει στην ημερήσια διάταξη την άμυνα της Ευρώπης σε μια στιγμή στην οποία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι ε, επεσήμανε και στους πολίτες και σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις ότι βρισκόμαστε ε, σε θέση να βελτιώσουμε τις δυνατότητες της άμυνας, γεγονός που έχει έμεσες ή άμεσες συνέπειες και στην άμυνα αλλά και στην ανταγωνιστικότητά μας και στη δυνατότητά μας για κοινοτομία. Και αυτή η διάσταση, η οποία είναι και στρατηγική και οικονομική, είναι στο επίκεντρο της συζήτησης που κάνουμε τώρα για την έρευνα. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ήταν λίγο πιο σαφείς ως προς την ανάγκη ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και η υπηρεσία μας να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για να δώσει κίνητρο για την ε, έρευνα και την καινοτομία. Επίσης το Συμβούλιο επενθύμησε ε, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια δράση για την έρευνα που σχετίζεται με την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στο γεγονό ότι η έρευνα για την υποστήριξη τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα υπάρχει με δύο βασικέ μορφέ. Καταρχάς, ε, έχουμε την έρευνα για τα προϊόντα διπλής χρήσης, τα οποία θα μπορούν να χρηματοδοτούνται από τα εφιστάμενα προγράμματα, όπως για παράδειγμα το ε, Horizon 2020, το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, και υπάρχει και μια διάσταση που θέλει να υποστηρίξει την εξωτερική πολιτική της Ένωσης σε θέματα ασφάλειας, την πρόληψη συγκρούσεων και τη διατήρηση της ειρήνης. Η δεύτερη μορφή έρευνας που είναι προς όφελος της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας είναι η έρευνα για την άμυνα που κάνουν τα κράτη-μέλη στα πλαίσια τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Έχουμε ένα αέρια ε, συστήματα, ε, θαλάσσια, χερσαία συστήματα και συστήματα πληροφορική και επικοινωνία. Κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες έχει μία λογική καινοτομία σε τη βάση ενός στρατηγικού θεματολογίου έρευνας ε, και δυνατότητα ανάπτυξης δυνατοτήτων. Okay. Thank you. Αυτό το σχέδιο ανάπτυξης των δυνατοτήτων έχει στόχο να βελτιώσει τις επιχειρησιακές ανάγκες που έχουν ε, προτεραιότητα οι ένοπλες δυνάμεις για την ανάπτυξη της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Τι μήνυμα λοιπόν ε, αποστέλλεται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για την έρευνα ε, που σχετίζεται με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Μας ζητήθηκαν να πάμε έτσι περαιτέρω και να δημιουργήσουμε μια νέα εργαλειοθήκη που θα είναι χρήσιμη για την άμυνα και θα είναι στην υπηρεσία της κοινοτομίας κάνοντας έκκληση να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που διαθέτει ο καθής. Καταρχάς ε, αυτά τα νέα εργαλεία. Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε κάτι το οποίο υπάρχει ήδη στο πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020 Θέλουμε αντιθέτως να δημιουργήσουμε ένα, ε, μοντέλο, ένα εργαλείο πληροφορικής το οποίο θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε τις δυνατότητες άμυνας για να υποστηρίξουμε τις μελλοντικέ επιχειρήσεις της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Αυτό, ε, τα εργαλεία θα πρέπει να έχουν συνέργειες με τα ε, εργαλεία έρευνας που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μπορέσει να βοηθήσει και την έρευνα η οποία στόχο έχει αυτή τη συνεργασία. Τώρα, τι είναι όλα αυτά τα οποία είναι χρήσιμα για την έρευνα. Θέλουμε να έχουμε μια πραγματική προστιθόμενη αξία στα, για την υποστήριξη των στοιχείων τα οποία χρειάζεται η Ευρώπη. Χρειαζόμαστε πράγματα τα οποία θα είναι σαφώς καθορισμένα και θα είναι διαρθρωμένα με βάση τις προτεραιότητες. Για παράδειγμα, ε, ε βάση των δυνατοτήτων που έχουμε για ασφάλεια και άμυνα, στα οποία σας ανέφερα προηγουμένως. Αναπτύσσοντας αυτές τις δυνατότητες λοιπόν που φαίνονται σε αυτό το σχέδιο ε, και που θα είναι στην υπηρεσία της κοινή πολιτικής ασφάλειας ε, και άμυνα στο σύνολό της η Ευρώπη θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει εξωτερικές κρίσεις παρά το γεγονός ότι έχουμε πολύ περιορισμένο προπολογισμό. Ε, το γεγονός ότι είναι ε, πολλαπλή αυτή η δυνατότητα είναι σημαντική. Δεν έχουμε μία προτεραιότητα αλλά πολλές προτεραιότητες που θα μπορεί να είναι χρήσιμοι και στις ε, ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις καθώς και στις πολιτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργαλεία στη διάθεση της καινοτομίας, τέλος. Θέλουμε να βρούμε τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες και να έχουμε σε και εδώ θέματα τα οποία έχουν ήδη εντοπίσει τα κράτη-μέλη και η βιομηχανία στα πλαίσια της ομάδας εργασίας που ασχολείται με τα θέματα αυτά σε τεχνολογικό επίπεδο. Όσον αφορά τη βιομηχανία, αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι και η δυνατότητά μας να καινοτομήσουμε, η ανταγωνιστικότητά μας και το ε, πώς μπορούμε να έχουμε τεχνολογικά και ε, στρατηγική σημασία στοιχεία για, στην υπηρεσία της κοινωνίας στις προπαρασκευαστικές δράσεις, στο κεφάλαιο για την στήριξη στη βιομηχανία και στην ανταγωνιστικότητα, υπάρχει μνήμα ε, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2013. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία από όλους τους φορείς. Καταρχάς, τα κράτη-μέλη, τα οποία ε, είναι αυτά τα οποία θα υλοποιήσουν την επιχειρησιακή διάσταση και θα κάνουν και τις κατάλληλες επιλογές ε, για τις ε, στρατιωτικές δυνατότητες οι οποίες θα θέσουν στην υπηρεσία της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι όλο και πιο ενημερωμένη για την τεχνολογία και τις καινοτομίες που θα πρέπει να κάνει μια πρόταση για μετά το 2016 ώστε οι προπαρασκευαστικές ε, δραστηριότητες να συνεχίσουν να υλοποιούνται μετά το 2017. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή υπηρεσία άμυνας που έχει μεγάλη πείρα στην επιλογή των τεχνολογικών προτεραιοτήτων, στην σε ε, επιχειρησιακές μας δυνατότητες και στην διεξαγωγή ε, περίπλοκων επιχειρήσεων που έχουν κυβερνητική, στρατιωτική διάσταση και βιομηχανική διάσταση. Και αυτό το οποίο μας λείπει είναι ο κατάλληλος προϋπολογισμός. Εδώ θα είμαι ειλικρινής. Αυτή τη δυνατότητα ε, αυτή τη στιγμή για να εντοπίσουμε τις, ε, ε, τους τομείς που θεωρούμε προτεραιότητες είναι πολύ μεγαλύτερες από τις πόρους που διαθέτουμε για να τα χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά. Η Φεντερίκα Μοναγκερίνη, η μελλοντική είπατε εκπρόσωπος εξωτερικών θεμάτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το στοιχείο αυτό και εγώ θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα να ε, συγκεκριμενοποιήσουμε το ρόλο της ασφάλειας και της άμυνας. Ε, και τέλος ο κλάδος, η βιομηχανία, η οποία θα είναι αυτή η οποία θα έχει τις πρώτες συνέπειες για αυτά τα θέματα ε, τα οποία αφορούν τη βιομηχανία και κυρίως τα πνευματικά δικαιώματα. Δεν καταλαβαίνω το συγκεκριμένο ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν. Ε, ορισμένες φορές μου φαίνεται ότι σας πιέζω ενώ εσείς είστε οι άνθρωποι που έχετε ήδη πιστεί για το ο γεγονός ότι πρέπει να υλοποιήσουμε τα θέματα αυτά. Υπάρχει και μια έκθεση της ε, ε, Επιτροπής σας η οποία ε, επιβεβαιώνει αυτό το γεγονός. Αναφέρομαι στην ανάγκη για νέες δράσεις, οι οποίες θα είναι χρήσιμες για την άμυνα της Ευρώπης και θα είναι και στην υπηρεσία της καινοτομία για τις προπαρασκευαστικές μας δράσεις. Αυτό ε, θα χρησιμοποιήσω και για τις δικές σας τις δράσεις, ε, για κάποια πολιτικά προγράμματα τα οποία έχουν προτείνει κάποιοι από εσά και που είχαν μεγάλη υποστήριξη στην Επιτροπή ΑΦΕΤ, στην Ήτρε και στην Επιτροπή Προπολογισμών ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ρόλο τον οποίο προβλέπετε για την υπηρεσία μας προς αυτό το σκοπό. Θα πρέπει να συγκλίνουν ε, ε, οι στόχοι των διαφόρων παραγόντων και να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί και ε, να υπάρχει και κάποια συγχρηματοδότηση και να υπάρχει συγχρηματοδότηση με κοινοτικού ε, και κυβερνητικού πόρου και να μην έχουμε μόνο ε, χρηματοδότηση για επιχειρησιακά στοιχεία αλλά και για τα υπόλοιπα. Και θα ήθελα λίγο να σα πω και λίγο πράγματα για όσου ε, χρηματοδοτούν. Θα πρέπει να έχουμε βέλτιστη χρήση των πόρων μα χωρί επικαλύψει και να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες συνέργειες και να χρησιμοποιούμε ό,τι εργαλεία διαθέτουμε στη διάθεσή μα. Εάν έχουμε και στρατιωτική ε, συνέργεια μεν, αλλά θέλουμε να έχουμε και ε, κοινοτική και διακυβερνητική συνεργασία και όλα αυτά σε στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό λοιπόν το οποίο επιθυμώ ως φορολογούμενος πολίτης είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση η οποία θα μας επιτρέψει κάθε ευρώ που επενδύεται να δίνεται για κατάλληλους ε, πόρους και να μην είναι ε, σε καμία περίπτωση δράση μας αντιπαραγωγική. Επιτρέψτε μου τώρα να σας μιλήσω για τη συνέχεια των παραπαρασκευαστικών δράσεων. Όπως το λέει και ο ίδιος ο όρος, οι προπαρασκευαστικές δράσεις είναι το πρώτο στάδιο. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει στη συνέχεια είναι το τι μέλη γενέστε. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό και η δημιουργία ενός κατάλληλου μέσου για την έρευνα που θα έχει και όλες τις πτυχές ε, της πολιτική πολιτικής ασφάλειας και άμενας συμπεριλαμβανομένης και της άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το σκοπό θα πρέπει οι προπαρασκευαστικές δράσεις να μας δώσουν απτά αποτελέσματα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουν να πείσουν για τη συνέχεια. Και θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι το σύνολο του βιομηχανικού κλάδου θα μπορεί να συμμετέχει. Να υπάρχει μεγάλη γεωγραφική ε, κάλυψη επίσης, κάτι το οποίο είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Και ε, η μέθοδος είναι εξίσου σημαντική με το περιεχόμενο σε αυτή την περίπτωση. Διότι η μέθοδος ε, είναι αυτή η οποία θα ξαναχρησιμοποιήσουμε για δράσεις μεγάλης κλίμακας στη συνέχεια. Όσον αφορά το περιεχόμενο τώρα, θα πρέπει να καθορίσουμε τις προτεραιότητές μας, να γίνουν μελέτες εφικτότητας και ε, να εξετάσουμε και τι υπάρχει σε τεχνολογικό επίπεδο και θα μας χρειαστεί και μία πληθώρα θεμάτων και εργαλείων τα οποία θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, για το στόχο μας. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να βεβαιωθούμε ότι η διαδικασία που θα προτείνουμε θα μας εγγυάται ότι το αποτέλεσμα θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές προτεραιότητες και τις ανάγκες ε, που έχουμε τώρα αλλά και στο μέλλον. Όσον αφορά τον τρόπο τώρα, επειδή είναι πολύ ευαίσθητα τα θέματα τα οποία συζητούμε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποια ουσιαστικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα, καταρχάς ε, τους κανόνες για την πνευματική ιδιοκτησία, που θα πρέπει να επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να μπορούν να εκμεταλλεύονται τα αποτελέσματα, και ταυτόχρονα να εγγυόμαστε ότι θα υπάρχουν και κίνητρα για τι επιχειρήσει. Δεύτερον, μηχανισμοί χρηματοδότησης μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης μεταξύ κρατών μελών και ε, τμήματος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλα αυτά τα θέματα θα συνδιοργανώσουμε ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σεμινάρια. Το πρώτο προβλέπεται για τις 21 Νοεμβρίου και θα ήθελα, ε, επειδή είναι εδώ ο κύριος ε, Ταρκάσκι, ε, το Κάρσκι, να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την εξαιρετική δουλειά που έγιναν από τις ομάδες μας που συνεργάστηκαν στενά. Προφανώς και ο κλάδος της βιομηχανίας θα συμμετέχει σε αυτά τα σεμινάρια, αλλά ε, θεωρώ ότι η συμμετοχή της Επιτροπής σας επίσης στις εργασίες που είναι μεν αρκετά προχωρημένες θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Ολοκληρώνοντα, θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστέ και πιο αποτελεσματικοί. Να μπορούμε να ε, ξεπεράσουμε τις ε, στήρες αντιπαραθέσει και να μπορέσουμε να καταφέρουμε να έχουμε κάποια πρόοδο. Να μπορέσουμε να ελοπίσουμε την εντολή του ε, Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2013, να ανταποκριθούμε στην έκκλησή σα για μεγαλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προετοιμάσουμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2015. Έτσι, η κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το ευμετάβλητο κλίμα που αντιμετωπίζουμε όλο ένα και περισσότερο. Και εδώ έρχομαι στην ανταλλαγή απόψεων που έγινε την περασμένη Τρίτη με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την οποία παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η άμυνα και η κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα ε, βεβαίω δεν γίνονται ανεξάρτητα από άλλες μορφές δράσης, αντιθέτως συνδέονται με τους στρατηγικούς μας στόχους και με τις δυνατότητες δράσης μας βάσει των αξιών μας και θέλουμε πάντα να έχουμε θετικέ συνέπειες σε θέματα καινοτομία και θέσεων αποσχόληση και να υπάρχει υψηλή προστιθέμενη αξία. Κάθε ευρώ που επενδύεται στην άμυνα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία. Και ελπίζω ότι η Επιτροπή σα, στη νέα τη σύνθεση θα συνεχίσει να μα οθεί, να δίνουμε σαφείς απαντήσει στις προκλήσει και σα ευχαριστώ πολύ που τίνατε στα όσα είχα να πω και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σα. Ευχαριστώ. Thank σας ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Σλαβό Μιλτοκάρσκι, προεστάμενο της Διοικητικής Μονάδας ε, της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων Βιομηχανίας ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Τοκάρσκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ κάποια στοιχεία, γιατί πολλά από τα ζητήματα παρουσιάστηκαν ήδη από τον προλήσαντα και είναι και απόδειξη άλλωστε αυτό της καλής μας συνεργασίας. Οπότε και τα μηνύματα που θέλουμε να αποστείλουμε είναι παρόμοια. Αλλά θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια για τις συνέργειες μεταξύ της ε, διπλής χρήσης έρευνας ε, για πολιτικούς και στρατιωτικούς σκοπούς και ε, ορισμένα ορόσημα που έχουμε θέσει όσον αφορά τις προβασκευαστικές εργασίες στο μέλλον. Να να πω για ποιο λόγο η Κομισιόν πρότεινε αυτές τις χρηστικές ε, εργασίες και έθεσε επιτάπητος την ε, μεγαλύτερη συνεργασία σε πολιτικά και στρατιωτικά ζητήματα στον τομέα της έρευνας. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όταν εξετάζουμε την λογική και την ε, χρησιμότητα. Ε, βεβαίως ο λόγος είναι ο μειούμενος προϋπολογισμός Επομένω, είχαμε την κατάσταση ε, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις στο μέλλον όσον αφορά την άμυνά τη, και να δημιουργήσει ε, μια, ε, την, το, το επαρκές το απαιτούμενο πλαίσιο για την έρευνα. Γι' αυτό για το 2014 η Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο δύο δράσεις και Είμαστε μεγάλοι, πολύ ικανοποιημένοι που υπάρχει υποστήριξη από τα δύο αυτά θεσμικά όργανα και μας δόθηκε η εντολή να τα υλοποιήσουμε σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Για να σας, να σας πω δύο λόγια για τις συνέργειες διπλής χρήσης. Η ευκαιρία που παρέχουν ε, αυτές οι συνέργειες είναι το, προέρχεται από το γεγονός ότι ε, η πολιτική και η στρατιωτική έρευνα ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό ταυτίζεται. 60% ε, μπορεί να ε, αφορά και τους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς σκοπούς. Γι' αυτό και θέλουμε συνέργειες και γι' αυτό γνωρίζετε ότι το Horizon 2020 έχει πολιτικό προσανατολισμό αλλά παρόλα αυτά ε, μέσω των συνεργειών μπορούν ε, να ε, υπάρξουν, υπάρξει έρευνα και στον τομέα της άμυνας και της αμυντικής οριμότητας. Αυτό που κάνουμε τώρα και το κάνουμε και στη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας είναι ότι κοιτάζουμε αυτές τις δυνατότητες διπλής χρήσης του Horizon 2020 και το στοιχείο που ε, είναι πιο κατάλληλο για διπλή χρήση έρευνα είναι η τεχνολογία και θα εξετάσουμε συγκεκριμένα ποια ε, προγράμματα, ποια έργα ε, θα είναι τα καταλληλότερα για τα επόμενα χρόνια και θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις συνέργειες που επιδιώκουμε. Πριν από δύο μέρες, την Παρασκευή, ε, δημοσιεύσαμε και ένα εγχειρίδιο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μεταξύ άλλων εξηγεί λεπτομερώς ε, τι είναι αυτά τα έργα dual use, διπλής χρήσης, πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν τα ερευνητικά προγράμματα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, αλλά και σε συνεργασία με διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Διαρθρωτικά ε, ε, ε ταμεία, το Horizon 2020 και νομίζουμε ότι με αυτό το εγχειρίδιο θα καταφέρουμε να διαδώσουμε αυτήν την, την ιδέα των έργων διπλής χρήσης που η δυνατότητα για αυτά υπήρχε βέβαια μέχρι τώρα, αλλά πολύ λίγες μικρομεσαίες επιχειρήσεις την αξιοποιούσαν. Θέλουμε δηλαδή με κάποιον τρόπο να ε, φέρουμε, ε, να αξιοποιήσουμε περισσότερο ε, αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την χρηματοδότηση ε, έργων διπλής χρήσης. Τώρα για τις προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως είπε και ο κύριος Ροζιέ, δεν μιλούμε αποκλειστικά για προπαρασκευαστικές εργασίες. Ε, αυτές μάλλον θα χρηματοδοτηθούν ε, με περιορισμένους πόρους. Αυτό που, μπορούμε να, ε, αυτό που αλλάζει είναι ότι στο επόμενο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο μπορούμε να έχουμε πλήρη έρευνα για ζητήματα κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Και από αυτή την άποψη πρέπει να εξετάσουμε και το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα της προκορασκευαστικής εργασίας. Επίσης, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ποια είναι, ποια είναι το πρόσθετο όφελος αυτής της ε, μελλοντική έρευνα σε επίπεδο ευρωπαϊκή. Νομίζω ότι μπορούμε να αναφέρουμε τουλάχιστον τρία στοιχεία που σχετίζονται με αυτή την προστιθέμενη αξία. Πρώτον, ε, η βιομηχανική ε, σκοπιά. Ελπίζουμε ότι μέσω της χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να ε, ενισχύσουμε την βιομηχανική συνεργασία, τη δημιουργία βιομηχανικών δικτύων και να δημιουργήσουμε εκείνη την κρίσιμη μάζα που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί. Και μέσω αυτής της, αυτού του είδους υποστήριξης που θα παρέχουμε μπορούμε να βοηθήσουμε και την βιομηχανία να διατηρήσει και να αναπτύξει παραπέρα εκείνες τις δυνατότητες ε, δράσης ή εκείνες τις βιομηχανικές ε, δυνατότητες που θα είναι ε, απαραίτητες στο μέλλον για να δημιουργηθούν δυνατότητες σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας που χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ακριβώς αυτές οι δυνατότητες σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Είδαμε στα τελευταία συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου ότι υπήρξε συμφωνία των κρατών μελών επί της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, ενδεχομένως να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες ε, στο μέλλον και αυτά τα ερευνητικά προγράμματα θα, δώσουν, θα μας δώσουν περισσότερα εργαλεία για την υλοποίηση της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Οπότε μιλάμε για μια έρευνα που σχετίζεται με τις δυνατότητες που στόχο έχει να αναπτυχθούν ακριβώς αυτές οι δυνατότητες που θα βοηθήσουν την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας της. Στο μέλλον επίσης ε, θα έχουμε και αυτό που ονομάζουμε ενισχυτή δυνατοτήτων. Ένας τρόπος δηλαδή που έχουμε για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να συνδυάσουν τα, τις δυνατότητες τους που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν διάσπαρτες. Δημιουργούμε δηλαδή μια πλατφόρμα ώστε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες και εδώ υπάρχει ήδη ένα παράδειγμα στη θαλάσσια ασφάλεια όπου ακριβώς υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών. Είναι ένα θετικό παράδειγμα δηλαδή ε, που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και ε, στο μέλλον. Τώρα να πω και δύο λόγια για το χρονοδιάγραμμα και ποια είναι τα βασικά ορόσημα που έχουμε μπροστά μας. Όπως γνωρίζετε η Επιτροπή έχει ε, αναπτύξει έναν οδικό χάρτη που υιοθετήθηκε φέτος τον Ιούνιο όπου συγκεκριμενοποιήσαμε λίγο τους τρόπους και τους επιδιωκόμενους στόχους και μετά από αυτά τα εργαστήρια σε συνεργασία με την Επιτροπή σας και τις συζητήσεις με τους διαφορούς ενδιαφορεωμένους θα προσπαθήσουμε να ε, φέρουμε μαζί, να, φέρουμε σε ένα, να, να γίνει συζήτηση μεταξύ κρατών μελών, της βιομηχανίας και του Κοινοβουλίου για να κατακτηθεί μια κοινή αντίληψη για το ποια, ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο της προγραμματικής εργασίας. Ιδανικά κατά τη γνώμη μας ε, θα θέλαμε να επιτευχθεί μια τέτοια πρόοδος ώστε ήδη τον Ιούνιο του 2015 να, σημειωθούν, να σημειωθεί στα, ευρωπαϊκά, στο, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2015. Πριν από λίγους μήνες, όταν είχα ε, έρθει ξανά εδώ, ανέφερα ότι η προθεσμία για την έναρξη των προπαρασκευαστικών εργασιών θα είναι το 2018. Στο μεσοδιάστημα συνεργαστήκαμε με τους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού και την Νομική Υπηρεσία και φαίνεται ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάτι τέτοιο και το 2017. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να επιδείξουμε, να παρουσιάσουμε αυτά τα σχέδια, τα έργα που έχουμε μπροστά μας ε, ώστε να μπορέσουν να ε, οριστικοποιηθούν και έγκαιρα κατά την συζήτηση του νέου δημοσιονομικού ε, πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί διαπιστώθηκε ότι αν ξεκινήσουμε το 2018 ενδεχομένως να μην έχουμε τον απαραίτητο χρόνο για να αποδείξουμε την αξία αυτής της ερευνητικής δουλειάς που θα γίνει στο μέλλον. Αν ξεκινήσουμε τώρα το 2017, σύμφωνα με τη δημοσιονομική διαδικασία, θα πρέπει να ε, παρουσιάσουμε ένα πρώτο προσχέδιο ε, της προπαρασκευαστικής, ε, των, των προπαρασκευαστικών εργασίων την Άνοιξη του 2016. Δεν είναι πολύ χρόνο. Ε, τι θα πρέπει να συζητήσουμε με όλους τους ενδιαφερόμενους και στις αρχές του 2016 δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσουμε ε, τη συζήτηση για αυτό το ζήτημα. Κάτι που θα μπορούσε να, να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016 και το 2017 να ξεκινήσουν οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως είπα. Νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ και βεβαίως ε, με πολύ μεγάλη χαρά θα απαντήσω στα ερωτήματά σας. Oh. Ευχαριστούμε, κύριοι, για αυτή τη συνοπτική παρουσίαση που μας κάνετε. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, επιτρέψτε μου να θέσω και εγώ δύο ερωτήματα και για τους δύο μιλητές. Πρώτον, για την πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία για αυτήν την διπλή χρήση που αναφέρατε της έρευνας που θα ενισχύσει έτσι τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσα στα πλαίσια ιδιαίτερα του ορίζοντα 2020. Πώς θα διασφαλιστεί η συνοχή όλων αυτών των στοιχείων. Πώς προβλέπετε να πετύχετε στην εφαρμογή των προπαρασκευαστικών δράσεων και πέρα από αυτά πώς θα χρησιμοποιηθεί ακριβώς το σύστημα της έρευνας γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστιες ανισότητες και διαφορές μεταξύ των παλαιών χωρών μελών και των νέων. Πώς θα διασφαλίσετε λοιπόν αυτή τη διάσταση της συνοχής. Δεύτερον, τα κριτήρια της συνεργασίας με τρίτες χώρες στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος. Και αναφέρομαι εδώ πάλι στη χρήση των ταμείων συνοχής που και των σχεδίων που έχουν κάποια σχέση με την ΚΠΑΣΑΜ γιατί και η εσωτερική και η εξωτερική συνεργασία μπορεί να κινητοποιηθεί με εξωτερικούς εταίρους Πώς θα τα δομήσετε όλα αυτά, με τι κριτήρια. Ο κύριος Όιλερ νομίζω θέλει να πάρει το λόγο τώρα. Θα τεθούν όλα τα ερωτήματα ή μάλλον ο πρώτος γύρος και μετά θα απαντήσουν οι ομιλητές. Ναι, καταρχάς κάτι που ανέφερε και η Πρόεδρος για τη συνοχή. Είναι σαφές ότι στον ορίζοντα 2020 δεν υπάρχει διάσταση συνοχής. Είναι το μόνο πρόγραμμα της Ένωσης όπου δεν παίζει ρόλο η συνοχή ακόμα. Στην πράξη όμως έχω δύο ερωτήματα αναλύοντας το πρόγραμμα 14-15 άμα κοιτάξετε καλά θα δείτε ότι τουλάχιστον έτσι όπως παρουσιάστηκε στο υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο είμαστε ακόμα στη φάση της επιτροπολογίας και έχουν ταυτιστεί τέσσερις στόχοι κυρίως μεταξύ των οποίων και η ψηφιακή ασφάλεια και άλλοι. Από συστηματική όμως απόψεως, ξέρω ότι είναι πολύ θεωρητικά αυτά που λέω, αλλά αυτά τα θέματα που εγκρίνατε αφορούν άλλου είδους αποστολές, όχι καθαρά της ΚΠΑΣΑΜΑ. Ας πούμε η ασφάλεια στα σύνορα ή η διαχείριση της πληροφόρησης για τις ανθρωπιστικές αποστολές που αναφέρεται εδώ ή η διαχείριση της πληροφόρησης για τις υποδομές των εξωτερικών δράσεων. Αυτά τα βρίσκω λίγο περίεργα γιατί τέτοια θέματα αφορούν κυρίως το συνδυασμό πολιτικής και στρατιωτικής δράσης. Γιατί αποκλείστηκε από όλα αυτά τα θέματα η στρατιωτική πτυχή. Δεν συμβαδίζει αυτό με αυτά που μας είπατε. Δεύτερο ερώτημα. Υπάρχει κάποια δομική διαφορά ή χάσμα Δηλαδή υπάρχει μια πτυχή βιομηχανικής πολιτικής και υπάρχει και μια άμεση σχέση με αποστολές της ΚΠΑΣΑΜ. Στο παρελθόν τα χρήματα αυτά προέρχονταν από την RGD και τώρα ο προϋπολογισμός που προβλέπεται και οι δομές θα χορηγούνται από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό, προβλέπει δηλαδή τελείως διαφορετική δομή. Ποια ήταν η πρόθεση της Κομισιόν, γιατί αυτά τα 1,7 δισεκατομμύρια πήγαν από τη μία Γενική Διεύθυνση στην άλλη, στην εσωτερικών δηλαδή. από τη μία υπάρχουν τα καθαρά θέματα της ΚΠΑΣΑΜ και από την άλλη τα βιομηχανικά. Αλλά ούτε το ένα ούτε το άλλο δεν είναι θέμα εσωτερικών. Γιατί τα αναθέσατε στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών. Ευχαριστώ κύριε Λούζινγκ. Θα μιλήσω στα γερμανικά. Κύριε Ροζιέ, είπατε ότι θα πρέπει να ε, μπούμε στη θέση του φορολογούμενου και βγάλατε το, συμπεράσμα, το συμπεράσμα, τα συμπεράσματά σας με βάση αυτή την προσήγγιση. Αν μπω εγώ στη θέση ενός φορολογούμενου, θα μπορούσα να φανταστώ για παράδειγμα ότι θα ήθελα Θα ήθελα να τηρηθούν οι διατάξεις της, ε, του άρθρου 42 παράγραφου, της παραγράφου 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγορεύει πολιτικές δράσεις με στρατιωτικά ε, μέσα. Γιατί αν κατάλαβα σωστά υπόθηκε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε εκτός πλησίου εννοείται και τέτοιου είδους ε, φραγμούς, ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε και ε, πέρα από τις, πέρα από συνθήκες. διότι συζητούμε τις δυνατότητες για την έρευνα στο ε, τομέα της ασφάλειας προκειμένου να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έρευνα στη συνέχεια. Ε, έγινε μνήμα στην ε, έρευνα, την πολιτική και τη στρατιωτική, ώστε να μπορέσουμε να τη συνδυάσουμε για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλους αυτούς τους φραγμούς. Εγώ ερμηνεύω κατά αυτόν τον τρόπο αυτά τα οποία μας λέτε. Θεωρώ ότι ε, θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτό το φράγμα από αυτά που άκουσα να λέτε. Και αναφέρομαι στην έκθεση της Επιτροπής για την Άμυνα την ετήσια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και ο κύριος Έουλερ αναφέρθηκε στις προπαρασκευαστικές δράσεις και νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση αναφερόμαστε ανοιχτά σε, αυτή την, ε, σε αυτόν τον προσανατολισμό να προωθήσουμε την έρευνα για στρατιωτικούς σκοπούς. Θα ήθελα λοιπόν να έχω μια σαφή απάντηση σε αυτή την ερώτηση και θα ήθελα πραγματικά να μου πείτε κατά πόσον επιθυμείτε σε αυτή την περίπτωση να μην γίνει σεβαστό το κριτήριο των συνθήκων, το οποίο δεν προβλέπει χρηματοδότηση προς αυτό το σκοπό. Αναφέρεται επίσης και μία ομάδα ε, προσώπων τα οποία θα συμμετέχουν ε, στην προετοιμασία αυτών των μέτρων. Στην τελευταία αυτή ομάδα προσωπικότητων ασκήθηκε κριτική ότι η σύνθεση αυτής της ομάδας ήταν πολύ μονόπλευρη. Πώς διασφαλίζεται λοιπόν ότι ε, ε, ε, η ομάδα αυτή αυτή τη φορά θα είναι κάπως πιο πλουραλιστική ως προς τη σύνθεση της και θα υπάρχουν και επικριτικοί της πολιτικής συμμετέχοντες. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, εγώ θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει τουλάχιστον σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπίσουμε για παράδειγμα ε, την κριτική που ασκείται για το γεγονός ότι η πολιτική μας χαράσεται υπό την πίεση των ε, λόμπι. Κύριε Μπάιος και στη συνέχεια ε, θα μπορούν να πάρουν το λόγο τα άλλα μέλη για να θέσουν τα ερωτήματά τους. Και εγώ παρόμοια ερωτήματα είχα. Στην ομάδα των Πρασίνων ε, είμαστε αντίθετοι με τη χρήση ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων για σκοπούς άμυνας και αυτό συμπεριλαμβάνει και την έρευνα για την άμυνα και υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο ένας είναι ότι θεωρούμε ότι δεν υπάρχει βάση δικαίου για τη χρήση τέτοιων κονδυλίων και πώς μπορεί κανείς να ορίσει αυτή την έρευνα σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, ποια είναι τα όρια. Και αν τελικά χρηματοδοτηθεί μια τέτοια έρευνα από ευρωπαϊκά κονδύλια, σε ποια γραμμή του προϋπολογισμού θα πιστοθούν ε, αυτά τα χρήματα. αν δεν χρηματοδοτηθούν ε, τα έργα αυτά στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020. Κύριε ε, Γκάλα, εσείς είχατε τον λόγο κανονικά. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ νωρίτερα, αλλά αυτή τη στιγμή η πρόεδρος λέει ότι εννοούσε ότι δεν του έδωσε το λόγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, ζητώ συγγνώμη γιατί ε, δεν ήμουν εδώ, διότι ήμουν στη συνεδρία συγκρότησης αντιπροσωπείας και είμαι πρόεδρος εκείνης της αντιπροσωπείας, οπότε ζητώ συγγνώμη. Μια ερώτηση για τον κύριο Ροζέ τονίσατε ότι στις προπαρασφαιστικές εργασίες είναι σημαντικό να διασφαλιστεί αυτό που θα ε, προκύψει. Τι περιμένουν λοιπόν τα κράτη-μέλη από αυτήν την έρευνα που σχετίζεται με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμενας που θα ξεκινήσει από το 2021 στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και μια ερώτηση προ την Κομισιόν αυτή βεβαίω. Κύριε Τοκάρσκι, εσείς είπατε Μιλήσατε για το ορίζοντα 2020 και την ε, πολιτική διάσταση, του, τον πολιτικό χαρακτήρα αυτού του ε, προγράμματος. Οπότε πώς μπορούμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα ε, σε σχέση με την στρατιωτική έρευνα. Υπάρχουν ε, λοιπόν συγκεκριμένες πολιτικές διαστάσεις του προγράμματος αυτού. Και θεωρώ ότι και εν μέρει απαντώ και ε, σε αυτό που είπε η συνάδελφος από τους, προς, Πρασίνους. Νομίζω ότι το όριο λοιπόν θα πρέπει να είναι ότι η έρευνα αυτή θα πρέπει να αποστηρίζει τις αποστολές στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Ασκούμε πολιτική που ε, ομόφωνα από τα κράτη-μέλη και με καταπλειοψηφία από το Κοινοβούλιο έχει εγκριθεί όταν κάνουμε τέτοιες αποστολές θα πρέπει βεβαίως να υποστηρίζουμε τους εαυτούς μας, να το πω έτσι, με ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν έχει κανένα νόημα εδώ πέρα με ένα σχιζοφρενικό τρόπο να παρουσιάζουμε μια εικόνα ότι από τη μία πλευρά είναι η καλή και από την άλλη πλευρά είναι η κακή. Ε, και η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας είναι μια ηθικά νομιμοποιημένη και καλή πολιτική. Δεν είναι ούτε ανήθικη ούτε κακή. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσει που έχουμε και στις ανάγκες μας. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι μπορούμε να αφιερώσουμε συγκεκριμένες πιστώσεις του προπολογισμού που θα κατευθύνονται σε αυτές τις αποστολές προκειμένου να χρηματοδοτούνται με συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αλλά θα ήθελα να ακούσω και την δική σας άποψη από αυτού του θέματος. Thank you. Maybe Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ροζέ ίσως πρώτα και μετά ο κύριος Τοκάρσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλά τα ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω με τη σειρά. Καταρχήν η πρόσβαση στα κοινωνικά ταμεία. Συνεργαστήκαμε πολύ με την Κομισιόν για να φανούν τα όρια της χρήσης των κοινωνικών ταμείων για τα διπλής κατευθύνσεως προγράμματα. Κανονικά δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα κοινωνικά ταμεία, αλλά από το κοινωνικό ταμείο. Αλλά συνεργαζόμαστε με όλα τα Υπουργεία που διαχειρίζονται χρήματα του κοινωνικού ταμείου σε όλες τις χώρες μέλη. Επιλέξαμε μερικά από αυτά τα προγράμματα και θελήσαμε να τα προωθήσουμε ώστε να γίνουν συμβατά με τους στόχους του κοινωνικού ταμείου και αποδείξαμε ότι είναι δυνατόν νομικά να χρηματοδοτηθούν μερικά τέτοια διπλά προγράμματα από το κοινωνικό ταμείο εφόσον πρόκειται για έρευνα. Αναφέρατε τώρα γενικότερα το πρόβλημα της συνοχής. Ας απαντήσει η Κομισιόν καλύτερα γι' αυτό. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι προσέχουμε πάρα πολύ τη γεωγραφική ισορροπία που δεν είναι πάντα εύκολο να επιτευχθεί. Προσέχουμε όμως ιδιαίτερα τα ενδιαφέροντα των χωρών μελών. Ξέρουμε ότι στις περισσότερες η αμυντική βιομηχανία είναι σε κακή κατάσταση, αλλά προσπαθούμε κάτι να κάνουμε για να προωθήσουμε τα κυριότερα προϊόντα τους. Επίσης, η έρευνα που έχει αναλυθεί ήδη για θέματα ΚΠΑΣΑΜ ε, έχει εξεταστεί δεόντως από την Κομισιόν και το κύριο θέμα είναι η χρήση των κοινοτικών κονδυλίων για ορισμένες δραστηριότητες της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Όπως σας είπα και πριν προσέχουμε ιδιαίτερα την άποψη του φορολογούμενου και το νομικό υπόβαθρο. Για μένα το άρθρο 42 είναι μια σίγουρη νομική βάση και φαντάζομαι ότι δεν το ξέρουν βέβαια όλοι οι φορολογούμενοι αλλά ας είμαστε ρεαλιστέ. Αν ερμηνεύσουμε αυστηρά το 42 μπορούμε τότε να καταργήσουμε το μισό περιεχόμενο του ορίζοντα 2020 γιατί εκεί υπάρχει ένα τριπλό επίπεδο χαμηλής τεχνολογίας και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο αγοράς είναι ανταγωνιστική διαγωνισμοί και προμήθειες. Δεν μου αρέσει εμένα ο όρος διπλή χρήση. Γιατί συχνά είναι πολλαπλού στόχου τα προγράμματα αυτά και όχι απλώς διπλού. Το σημαντικό βέβαια για την έρευνα είναι να έχει ως το δυνατόν μεγαλύτερη οικονομική επίπτωση και αποτέλεσμα. Σήμερα έχει ισχύσει ένας συμβιβασμός που προβλέπει ότι υπάρχουν μερικές δυνατότητες για διπλή χρήση αλλά καμία δυνατότητα για χρήση προγραμμάτων ε, άμυνας και ασφάλειας στα πλαίσια του ορίζοντα 2020. Κατ' εμένα αυτό είναι ένα όριο που δεν ωφέλει την οικονομία. Και ξανάρχομαι στο, στην άποψη του φορολογούμενου. Υπάρχουν και νομικά όρια και φραγμοί, αλλά ας μην υπησύρθω σε αυτά. Υπάρχει το άρθρο 19 πάντως στον κανονισμό του ορίζοντα 2020, που λέει ότι πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε πολιτικά προγράμματα. Αν όμως με ρωτήσετε αν θα ήταν καλό να αλλάξει κάτι τέτοιο τότε θα έλεγα ότι εάν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε όσο δυνατόν περισσότερο το κάθε ευρώ του φορολογούμενου μέσα στα πλαίσια αυτής της δημοσιονομικής κρίσης βέβαια τότε θα απαντούσα ναι μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη εκμετάλλευση των συνεργειών και της συνεργασίας μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών προγραμμάτων. Τελευταίο ερώτημα του κυρίου Γκαλέ. Οι προσδοκίες μας για τη συνέχεια. Μόνο πρακτικά μπορώ να απαντήσω βλέπω, αναφέροντας τι βλέπω κάθε μέρα. Βλέπω ότι είναι πολύ ευκολότερο να υπάρξει ενδιαφέρον παρά χρηματοδότηση. Και το είχα πει και προηγουμένως, πιστεύω ότι η καταλληλότητα μιας διαδικασίας για να ταυτίσει προτεραιότητες που να υποστηρίζονται από πολλές χώρες μέλη είναι πολύ ψηλότερη από τη δυνατότητά της να βρει χρηματοδότηση για αυτές τις τεχνολογίες. Το πολύ ενδιαφέρον και το είπα και αυτό πριν είναι ότι όταν εξετάσουμε τις προτεραιότητες που προκύπτουν από την τελευταία ενημέρωση του προγράμματος βλέπουμε ότι μιλώντας για τις πραγματικές δυνατότητες βέβαια ότι η διπλή χρήση υπάρχει παραδείγματο χάρη για το Intertheater Airlift την αποστολή δηλαδή ανθρωπιστικής βοήθειας ή τροφίμων αεροπορικός υπάρχει δυνατότητα διπλής χρησιμοποίησης ή για το θέμα της προστασίας τα της χρήσης εκρηκτικών από πολίτες. Όλα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στρατιωτικά και πολιτικά στα πλαίσια της ΚΠΑΣΑΜ. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι το κύριο θέμα. Το κύριο θέμα για τα κράτη-μέλη είναι το εξή. Αν κάποια μέρα ξεπεραστεί το πολιτικό όριο, αν μας ζητήσουν να κάνουμε κάτι πραγματικά αποτελεσματικό στην ΚΠΑΣΑΜ, θα μπορούμε να το κάνουμε. Σήμερα όχι, αλλά αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Για μένα λοιπόν αυτό είναι το ερώτημα. Θέλουμε να δώσουμε στον εαυτό μας τα μέσα για μια πραγματική εξωτερική δράση. Ό,τι η φύση και να είναι η δράση αυτή. Αυτό είναι το ερώτημα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Στοκάρκη παρακαλώ. για την ερώτησή σας όσον αφορά τη συνοχή, την οποία όπως αντιλαμβάνομαι διατυπώσατε ε, όσον αφορά τη συνοχή της βιομηχανικής βάσης της άμυνας. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή εδώ. Αυτή η πολιτική αντανακλά την πραγματικότητα και αυτό είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα κάθε κράτος μέλος θέλει να διατηρήσει κάποιο τμήμα της αμυντικής της βάσης και υπάρχουν και κάποια κράτη-μέλη ε, στα οποία η βιομηχανική αυτή βάση είναι πιο ανταγωνιστική και υπάρχει ε, μία ανησυχία ότι αν όλα αυτά τα αφήσαμε στις δυνάμεις της αγοράς τότε μπορεί να υπάρχει μία μείωση της βιομηχανικής βάσης άμυνας που έχουν κάποια κράτη-μέλη. Και αυτό φυσικά ε, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, μεν είναι περιορισμένε οι δυνατότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά η διπλή χρήση από τα διορθωτικά ταμεία μα ε, προσφέρει τη δυνατότητα να δώσουμε μια απάντηση. Υπάρχει και μια καλή αμυντική βάση σε κάποια νέα κρατημέλη, αλλά όχι σε όλα. Και κάπω θα πρέπει να μπορούμε να αντισταθμίσουμε και τι επιπτώσει του ορίζοντα 2020 που βασίζονται στην αριστεία. Ταυτόχρονα είμαστε σε θέση να ε, σχεδιάσουμε τις προπαρασκευαστικές δράσεις κατά τρόπον ώστε τα κράτη-μέλη που η βιομηχανική βάση άμυνας τους υστερεί, να μπορούν να ληφθούν υπόψη και να μπορέσουν να έχουν κάποια νέα εξειδικευσή, όχι ανάπτυξη νέων συστημάτων, αλλά ίσως υποσυστημάτων. Εάν λοιπόν θέλετε να έχετε τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών για την προπαρασκευαστική δράση και το περιεχόμενό της, πρέπει να λάβουμε και αυτές τις πτυχές ε, υπόψη γιατί χρειαζόμαστε ομοφωνία. Δεν γνωρίζω την απάντηση για την πολιτική, ε, η οποία περιλαμβάνει, αν δεν κάνω λάθος, και την πολιτική συνοχή προς τρίτες χώρες. Συνοχή μεν προς τρίτες χώρες, αλλά μέσω προγραμμάτων, λέει η Πρόεδρος. Ναι, αναφέρθηκα στις τρίτες χώρες πρόγραμμα, ε, προγράμματα για έρευνα για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ε, σε συνεργασία με τρίτες χώρες ή δυνατόν. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί με τα κράτη-μέλη και αν μου επιτρέπετε θα είναι και ένα καθόδε ζήτημα. Δεν έχω κάποια απάντηση να σας δώσω αυτή τη στιγμή. σημειώνουμε ότι κάποια μπορεί να έχουν ε, πρόβλημα με την συμμετοχή τρίτων χωρών ε, ή κάποιων τρίτων χωρών στον ορίζοντα 2020. Δεν θα πω τίποτα άλλο γιατί ε, αυτό απαιτεί πολλές συζητήσεις και πολύ μεγάλο συντονισμό προκειμένου να υπάρξει κάποια συμφωνία. Όσον αφορά την ασφάλεια, νομίζω ότι η παρατήρησή σας ότι, που αφορά το πρόγραμμα ε, είναι κάτι το οποίο θα σας απαντήσω αργότερα. Ε, θα συμβουλευτώ και τους συναδέλφους, δεν μπορώ να μιλήσω εξ αυτών. Είναι κάτι το οποίο αποφάσισε τελικώς ο, ο κύριος Γιούνκερ. Η ασφάλεια θα περάσει στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και δεν μπορώ εγώ να το σχολιάσω αυτό. Και ε, είναι και κάποιο από τους λόγους τουλάχιστον για δύο θέματα, τη θαλάσσια ασφάλεια και την άμυνα στον κυβερνοχώρο, ε, ήταν το σκεπτικό να εξορθολογήσουμε λίγο τη δράση των διαφόρων γενικών διευθύνσεων και να υπάρχει και συντονισμός ε, ε, των ε, γενικών διευθύνσεων, στον οποίο θα ήταν σημαντικό να συντονίσει τα πράγματα κυρία Μογκερίνη. Αυτά είναι βέβαια προσωπική μου άποψη, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Γι' αυτό. Τώρα, για τον τίτλο, τη γραμμή του προπολογισμού για την προπαρασκευαστική δράση, να σας πω ότι εδώ είναι μια απλή διαδικασία προπολογισμού, αποφασίζεται μια ξεχωριστή γραμμή προπολογισμού και εδώ αναφέρομαι στις συγκεκριμένε δημοσιονομικές ε, προπτικές, γιατί θα ξεκινήσει η γραμμή προπολογισμού σε αυτές τις δημοσιονομικές προπτικές. Για το μέλλον, όντως, η πρόθεση είναι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και η σχετική έρευνα να βρίσκεται στο μελλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε δεκτό από τα κράτη-μέλη και την έχουν εγκρίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ε, θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει κάποια ε, αντίθεση με τις ε, συνθήκες και με αυτά τα οποία θα προτείνουμε εμείς. Όσον αφορά την ομάδα προσωπικότητων, εγώ να σας πω και πάλι ότι επειδή τώρα θα αναλάβει καθήκοντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαφίεται στον Επίτροπο να δει πώς θέλει, στην Επίτροπο μάλλον, να δει πώς θα θέλει να προχωρήσει το θέμα. Η αρχική πρόθεση ήταν να συσταθεί αυτή η ομάδα, ακολουθώντας ε, το παράδειγμα της προπαρασκευαστικής δράσης για την ασφάλεια και είχαμε και κάποιες ενδείξεις από κάποια κράτη-μέλη ότι θα ήθελαν η ομάδα αυτή να είναι λίγο πιο ε, ε, μεικτή, αν μου επιτρέπετε, να μην έχουμε μόνο στρατηγούς εκεί. Αυτό βέβαια θα το αποφασίσει η Επίτροπος αφόσον αναλάβει καθήκοντα και είναι ένα από τα πρώτα θέματα τα οποία θα τις θέσουμε και θα αποφασίσει η ίδια πώς ε, ε, θα προχωρήσει η διαδικασία και ποιος ίσως θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτή την ομάδα εάν υπάρχει ομάδα. Νομίζω ότι η τελευταία ερώτηση αφορούσε το πολιτικό σκέλος του ορίζοντα 2020 και το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, όπως σας είπα και προηγουμένως, εξετάζουμε ε, τους, ε, key enabling, τις Key Enabling Technologies, τις KETS, γιατί υπήρξε και μια σχετική μελέτη που προσπαθούσε να εξετάσει ποιοι τομείς ε, καινοτομία θα μπορούσαν να είναι σημαντικοί για τη βιομηχανία στο μέλλον. Και ένα τμήμα της μελέτης ε, αφορούσε την αμυντική κοινότητα και να δούμε πώς θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον ε, σε αυτούς τους τομείς και ε, από ό,τι φάνηκε υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και θέλουμε λίγο να το προχωρήσουμε αυτό διότι φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις ακόμα και όταν ασχολούνται αμυγός με πολιτική άμυνα ε, μπορεί να έχουν έρευνα η οποία θα έχει μεγαλύτερη σχέση με την άμυνα και κάποια άλλη όχι αλλά τμήμα του κόστους θα μπορούσε ίσως να προκύψει από τον ορίζοντα 2020. Ε, πρόκειται και για έρευνα ε, η οποία είναι χρήσιμη για πολλούς ε, τομείς και ίσως θα μπορούσε να συνεχιστεί και εκτός του ορίζοντα 2020. Έχουμε κάποια παραδείγματα στην οποία συμμετείχε και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες πρακτικές εφαρμογές, να έχουμε και καλύτερη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων. Λοιπόν, θα γίνει ένας δεύτερος γύρος ερωτήσεων και εγώ θα ήθελα να ε, μπούμε στο θέμα της ε, συνοχής. Ε, εγώ μιλούσα για τις διαφορές όχι μόνο εντός της αμυντικής βιομηχανίας αλλά και όσον αφορά τη δύναμη των ερευνητικών Ινστιτούτων. Αυτό που, ήταν, ε, το, αυτό που ρώτησα είναι ποιο, πώς οραματίζεστε όλο αυτό το δίκτυο ερευνητικών ιδρυμάτων. Κατανοώ ότι υπάρχει ένα πακέτο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ε, σε πολλές χώρες υπάρχει τεχνολογική πρόοδος και γνώση. Αυτό είναι προφανές αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και μεγάλα ερευνητικά Ινστιτούτα που έχουν πολύ συγκεκριμένες δυνατότητες να παρέχουν ε, τεχνογνωσία. Οπότε, ποιο είναι το σχέδιο εδαφικής ε, κατανομής και ποιο είναι το σχέδιο όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ αυτών των Ινστιτούτων. Ξέρω ότι οι Γερμανοί κάνουν μαθήματα και δεν είναι πολύ καλό αυτό, αλλά μιας και ήμουν εγώ ε, ο εισηγητής θα μπορούσα ίσως να διευκρινίσω ότι βασιζόμαστε στις βασικές αρχές του Horizon και το Horizon είναι το μόνο τμήμα του προϋπολογισμού που δεν ε, ε, σχετίζεται με τη συνοχή. Αφορά μόνο την, την έρευνα και την αριστεία. Αυτό που προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε στο πρόγραμμα και αφορά βεβαίως και στα ε, ερευνητικά προγράμματα για την άμυνα είναι η διεύρυνση της συνεργασίας. Είναι ένα πρόγραμμα που εξυπηρετεί και αυτόν τον σκοπό, αλλά επί της αρχής είναι μεταξύ των ελάχιστων γραμμών του προϋπολογισμού που δεν έχουν καμία σχέση με τη συνοχή, αλλά ο μόνος σκοπός είναι η αριστεία. Να επανέλθω και στο αρχικό μου ερώτημα. Νομίζω ότι η συζήτηση είναι κάπως παραπλανητική. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της αμυντικής έρευνας και η απάντηση είναι σαφής. Δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την αμυντική έρευνα στο πλαίσιο του Horizon 2020. Ταυτοχρόνως όμως υπάρχει σαφής ε, ε, κατεύθυνση ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, εργαλεία αλλά επειδή είναι λίγο επικίνδυνη αυτή η χρήση της ορολογίας θα ήθελα να, να χρησιμοποιήσω εγώ τον όρο της, ε, ε, των τεχνολογιών γεφύρωσης. Αυτό που, αυτό βρίσκεται πίσω από την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, από το γεγονός ότι επικεντρωθήκαμε σε αυτήν την πολιτική, είναι το εξής. Παρά το γεγονός ότι είναι μεγάλο το ερευνητικό πεδίο και πολύ λίγος ο, πολύ λίγα τα κονδύλια του προϋπολογισμού, επικεντρωνόμαστε στις αποστολές. Για παράδειγμα στη Λιβύη δεν υπήρχε καμία υποστήριξη σε άλλες αποστολές δεν υπήρξε δυνατότητα επικοινωνία μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών ε, ομάδων, το οποίο επίσης δημιουργεί κινδύνους. Και στη Συρία θα υπάρξει υποστήριξη μη στρατιωτικών αποστολών, διότι σε διαφορετική περίπτωση ε, μπορεί να δημιουργηθούν μεγάλοι κίνδυνοι ε, για τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτέ τι επιστολές, αυτές τις αποστολές. Αυτή ήταν λοιπόν η πρόθεση. Και αυτό είναι και το ερώτημά μου που δεν έχει απαντηθεί μέχρι στιγμής. Όταν σκέφτομαι πώς ορίζεται αυτή τη στιγμή το πακέτο αποστολών κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον λέγεται ότι θα δοθούν 350 εκατομμύρια ευρώ. Πρακτικά όμως μόλις 7 ή 5% αυτού του πακέτου όπως περιγράφεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής θα κατευθυνθεί στις αποστολές και ακόμη πιο πρακτικά, αν έτσι γίνουν τα πράγματα, στη γραμμή προϋπολογισμού για τα, για τα σύνορα, για παράδειγμα, υπάρχει ε, πίστοση για την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά δεν αναφέρεται καθόλου ότι αυτή αυτό το, αυτή η γραμμή έχει πολιτικο-στρατιωτική διάσταση, διότι διαφορετικά δεν θα μπορούσε να, να εφαρμοστεί καν. Οπότε, Πώς ακριβώς συνδέονται όλα αυτά με τη διάσταση της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Και αυτό το ζήτημα συζητήθηκε εκτενώς και σαφώς γιατί δεν υπάρχουν ακόμη ε, ισχυρές ενδείξεις ότι σε, αυτές τις, σε αυτά τα 350 εκατομμύρια περιλαμβάνονται και οι αποστολές. Και θυμίζω ότι είχε υπάρξει ευρία συνένεση για το γεγονός ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να κατευθυνθούν στις αποστολές. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κύριε Μπάρης. Yes, Ναι, έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Ροζέα, διότι είπατε, αν κατάλαβα καλά, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και οι οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έρευνα διπλής χρήσης. Διότι προηγουμένως ρώτησα πού τίθεται και το όριο. Το όριο που θα χρησιμοποιήσετε ποιο είναι. Ο κύριος Έλερ είπε ότι δεν θέλει να τα αποκαλεί διπλή χρήση και είπε ότι θέλει να τις λέει bridging technologies, τεχνολογίες που γεφυρώνουν. Ε, καταλαβαίνετε βεβαίως ότι υπάρχουν περιορισμοί στη διπλή χρήση, διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, στον πόλεμο, σε επιχειρήσεις ε, πολεμικής και να επανέλθω και στο θέμα των φορολογουμένων, διότι δεν θεωρώ ότι οι φορολογούμενοι θέλουν να χρηματοδοτήσουν παραγωγή ή έρευνα η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά του λαού μιας άλλης χώρας ή σε μια ενόπλη σύραξη και ούτω καθεξής. Επομένως, οι φορολογούμενοι δεν ε, ε, ενδιαφέρονται μόνο για τα χρήματα τα οποία μπορεί να λάβει ο κλάδος και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Υπάρχει και το ηθικό ζήτημα. Δεν είμαστε ανόητοι οι φορολογούμενοι. Κύριε Ροζέχ. Α, συγγνώμη. Ο κύριος Πανστρεύσκη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα κάνω την ερώτησή μου στα πολωνικά. Καταρχάς, να σας πω ότι εκπροσωπώ μια άλλη ομάδα σε σχέση με τη συνάδελφο φορολογουμένων πολιτών και οι δικοί μου φορολογούμενοι πολίτες θα ήθελε να αυξηθεί η χρηματοδότηση της έρευνας υπέρ της άμυνας για στρατιωτικούς σκοπούς, διότι γνωρίζουν ότι η έρευνα αυτή είναι και στην υπηρεσία της πολιτικής προστασίας και στις στρατιωτικές αποστολές ε, χρησιμοποιούνται ε, κονδύλια για την έρευνα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια και για ειρηνικούς σκοπούς. Καταρχάς, υπάρχουν λύσεις για να μην χαθεί η χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο, να μην χάσουμε τις εθνικές λύσεις. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις ε, προκειμένου να μην είναι πολύ μεγάλες οι περικοπές. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες ώστε οι δαπάνες αυτές οι οποίες ε, προβλέπονται ε, για τις δημοσιονομικές προπτικές αυτές να προστατεύονται από κάποια υπερβολική περικοπή, ακόμα και φορολογικής φύσεως. Ε, επόμενη ερώτηση. Αναφερθήκαμε και στο νέο Ινστιτούτο για Νέες Τεχνολογίες, αλλά δεν συζητήθηκε και αυτή η προοπτική χρηματοδότησης, αλλά μια άλλη προοπτική χρηματοδότησης. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν πώς θα συντονιστούν οι διάφορες επιτροπές, ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις και να είναι πιο αποτελεσματικό το έργο τους, να μην υπάρχει μια κατάσταση στην οποία να υπάρχουν αμφιβολίες για τον καλό συντονισμό μεταξύ των υφιστάμενων συστημάτων. Η κυρία Σλόζιν. Θα μιλήσω γερμανικά, αν μπορώ. Πραγματικά εκπλήσωμαι από την συζήτηση εδώ. Ο κύριος Έουλερ μας είπε ότι αν παραγνωρίσουμε τους κανόνες διπλής χρήσης ε, θα καταλήξουμε στη φυλακή. Ε, ουσιαστικά δηλαδή επινοούμε έναν άλλον ορισμό για να συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Και αυτό πραγματικά με εκπλήσει. Ε, αυτή η αξιολόγηση των πραγμάτων είναι πολύ ε, ε περίεργη για μένα. Και μια ερώτηση για τον κύριο Γκάλερ, είναι εδώ. Ναι, εδώ είστε. Εγώ δεν είμαι νομικός, και δεν είμαι σε θέση να ερμηνεύσω ε, απόλυτα ό,τι λέει η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε κύριε Γκάλερ και δεν το έγραψα μεν, αλλά γι' αυτό και σας κάνω την ερώτηση. Εσείς είπατε ότι είμαστε δεοντολογικά από τη σωστή πλευρά. Ναι, αυτό είπατε. Χρησιμοποιήστε τον όρο ηθικός, δεοντολογικός. Εντάξει, ηθικό, όχι λογικό. Είμαστε λοιπόν από την ηθική σκοπιά εντάξει. Και αυτό μα δίνει το δικαίωμα να ερμηνεύουμε όπω επιθυμούμε. Αυτό εννοούσατε με αυτό που είπατε. Επομένως, αυτό το οποίο λέει το άρθρο 42.2 των συνθήκων δεν αμφισβητείται. Είναι θέμα ερμηνείας τι, πώς θα πρέπει να το ερμηνεύσω εγώ. Για μένα η ερμηνεία θα μπορούσε να είναι ότι η πλειοψηφία είναι από τη σωστή πλευρά της πλάστικας και ε, χρειαζόμαστε όμως και κάτι ε, για να υπερασπιστούμε αυτούς σε περίπτωση που αλλάξουν οι ισορροπίες. Και πραγματικά με εξέπλεξε η παρατήρησή σας αναφερθήκατε σε ερμηνεία του τι επιθυμούν οι φορολογούμενοι. Υπάρχει κάποιος ο οποίος ισχυρίζεται ότι οι φορολογούμενοι θέλουν λιγότερες στρατιωτικές παρεμβάσεις και κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι χρειάζονται περισσότερες στρατιωτικές παρεμβάσεις. Αλλά δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε τις συνθήκες ούτε κατά αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να βλέπουμε τι λένε οι συνθήκες. Αν δεν μας αρέσει, τότε θα πρέπει κάτι να κάνουμε προκειμένου να αλλάξουμε τις συνθήκες. Ελπίζω λοιπόν να μην υπάρξει η πλειοψηφία που θέλει να τις τροποποιήσει, αλλά αν υπάρχει τότε θα πρέπει και να γίνει. Όπως ε, είπε ο κύριος Γκάλερ, είπε και ο κύριος Έουλερ ότι οι πολιτικές αποστολές χρειάζονται και στρατιωτική υποστήριξη. Και γι' αυτό, ακριβώς το λόγο θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την ε, στρατιωτική έρευνη από τον προπολογισμό για τις ε, πολιτικές αποστολές, γιατί τα δύο θέματα είναι αλληλένδετα. Άρα χρειαζόμαστε μια διαφορετική ερμηνεία αν δεν ισχύει αυτό. Εγώ τουλάχιστον σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξα. Αυτό αντιλήφθηκα ότι λέγαμε. Και η ερώτησή μου είναι πώς ερμηνεύονται οι συνθήκες. Τι θέλει να κάνει η πλειοψηφία των ε, βουλευτών προκειμένου να ερμηνεύσει ε, τις συνθήκες όπως την εξυπηρετούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. θα ήθελα να ζητήσω από τους ε, κυρίους Ροζέ και Ταρκάσκη να απαντήσουν όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις Υπάρχει και μια πολιτική συζήτηση και δεν θέλω να παρέμβω εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, οπότε θα επικεντρωθώ μόνο στο, στα, στα γεγονότα και στα στοιχεία. Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ε, ταμεία, στον ορίζοντα 2020 υπάρχουν ε, ε, συγκεκριμένα, συγκεκριμένα κονδύλια. Ε, μου αρέσει αυτός ο όρος της ε, γεφύρωσης ή των πολλαπλών χρήσεων, ναι, εφόσον εξυπηρετούνται πολιτικοί στόχοι. Και αν πάμε λίγο παραπέρα, αν αρνηθούμε έργο που ίσως κάποια στιγμή θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι και στρατιωτικού ενδιαφέροντας, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε και την διακοπή της χρηματοδότησης διαφόρων έργων που χρηματοδοτούνται αυτή τη στιγμή από το διαρθρωτικό από τα διαφορετικά ταμεία. Για μένα είναι πιθανό να χρηματοδοτηθούν έργα που έχουν πολιτικό ενδιαφέρον. Βεβαίως με αυστηρή τήρηση των κανόνων. Όσον αφορά τις ερωτήσεις για τα φορολογικά κίνητρα δεν, είναι ζήτημα με το οποίο ασχολούμαστε εμείς. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τις δημοσιονομικές αρχές, τις φορολογικές αρχές, για να δούμε αν συνεργατικά ερευνητικά προγράμματα θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την απαλλαγή ΦΠΑ, για παράδειγμα ε, που θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για την ενίσχυση της συνεργασίας στο τομέα της έρευνας. Είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα ναι το πώ θα μπορέσουμε να δώσουμε δηλαδή φορολογικά κίνητρα για να ενισχύσουμε την ε, συνεργασία στον τομέα της έρευνας ε, σε διάφορους τομεί. Όσον αφορά την ερμηνεία των συνθήκων, δεν είμαι νομικός και δεν πρόκειται να σας δώσω συμβουλές για το πώς θα ερμηνεύσουμε τις συνθήκες. Όμως το μόνο που βλέπω εγώ όταν ε, εξετάζω συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι ότι υπάρχει ανάγκη κάποια ερμηνεία σε συγκεκριμένους τομεί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από λίγους μήνες ε, έγινε μια συζήτηση για το Κοπέρνικου. το πρόγραμμα για, την, ε, τη δορυφορική παρακολούθηση της γης. Αν θα μπορούσαν δηλαδή κάποιες εικόνες να χρησιμοποιηθούν και από, την, ε, από τους δορυφόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε συζήτηση και αποφασίστηκε ότι ναι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέτοιες εικόνες, σε πολύ μικρό ποσοστό βεβαίως, ε, σε σχέση με το συνολικό όγκο εικόνων του Κοπέρνικους, σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα πλέον και αυτή η δυνατότητα είναι πολύ χρήσιμα, χρήσιμη για πολιτικές αποστολές στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας για παράδειγμα μετά από φυσικές καταστροφές. Εδώ υπήρξε ένας συμβιβασμός και υπήρξε και κάποια ερμηνεία ε, των συνθήκων και του δευτερογενούς του παράγωγου δικαίου ε, όσον αφορά το ποιο είναι ακριβώς το όριο μεταξύ της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και τι βρίσκεται στο περιθώριο των δράσεων της ε, κοινότητας. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα ε, γι' αυτό. Η εντύπωσή μου πάντως είναι ότι ακόμη και χωρίς να αλλάξουμε τις συνθήκες και τηρώντας αυστηρά τις συνθήκες αυτές υπάρχει ακόμα περιθώριο για καλύτερη αξιοποίηση ε, κονδυλίων στο πλαίσιο της, ε, των ε, πολιτικών συνεργειών. Ο κύριος Στοκάρσκι, νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο κύριος Ροζιέ. Όταν μιλούμε για διαρθρωτικά ταμεία Πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά ε, έργα που είναι διπλής χρήσης. Μιλάμε για ημιαγωγούς, για αεροναυτιλία. Όταν, αν, πάτε σε μια έκθεση του, του κλάδου για παράδειγμα ε, μπορείτε να δείτε πάρα πολλές νέες τεχνολογικές καινοτομίες οι οποίες είναι διπλής χρήσης. Και πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε ποια ακριβώς χρήση θα έχει μια τεχνολογική εξέλιξη στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο μέλλον των λεχθέντων, αυτό που πρέπει εμείς να διασφαλίσουμε είναι ότι θα πρέπει να συμμορφώνονται τα έργα με τις προϋποθέσεις των διορθωτικών ταμείων. Να δημιουργούνται θέσει απασχόληση, να ενισχύεται η ανάπτυξη, γιατί σε τελική ανάλυση τα κράτη-μέλη είναι αυτά που ξοδεύουν αυτά τα χρήματα. Οπότε εκείνα θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τέτοιου είδου ε, ευθύνε, αρμοδιότητε. Για την ε, ε, ερώτηση όσον αφορά τα ωφέλη δεν έχω απάντηση, θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου. Για τον ορίζοντα 2020 και την έρευνα. Βασικός επιδιωκόμενος στόχος είναι η αριστεία και ένας από τους κανόνες χρηματοδότησης, ε, όλοι οι κανόνες χρηματοδότησης θα πρέπει να τηρούνται και με βάση αυτά θα πρέπει δηλαδή να υπάρξουν να με όλα τα κράτη-μέλη για να δούμε πώς μπορούν να ληφθούν και ε, υπόψη στη διαδικασία αυτή και οι απόψει τους. Όμως είναι σημαντικό ότι στην ανακοίνωση που προτείναμε αυτήν την σειρά ε, εργαλείων Σκοπός μας ήταν να διευκολύνουμε και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και αυτή η συνεργασία κρατών, το μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να αφορά και τον τομέα της έρευνας και εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια εργαλειοθήκη που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερες συνεργασίες, περισσότερες συνεργασίες μεταξύ κρατών μελών. για να ξεπεράσουμε και του, τα, ε, τους περιορισμούς, τα όρια μεταξύ παλιών και νέων κρατών μελών, για παράδειγμα. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό το, ε, για αυτό το ερώτημα για, την, ε, για το Ινστιτούτο Νέων Τεχνολογιών. Ρωτάτε αν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των γενικών διευθύνσεων και αν δεν θα υπάρξει διπλή χρηματοδότηση. Κανονικά η Κομισιόν όταν υπάρχει χρηματοδότηση προσπαθεί να δημοσιεύει έγγραφα που, θα, ε, που εξηγούν ποια ακριβώς είναι η αλληλεπίδραση, ο συσχετισμός μεταξύ των διαφόρων εργαλείων. Για παράδειγμα πρόσφατα δημοσιεύσαμε ένα έγγραφο με το οποίο εξηγούμε πώς το Horizon 2020 θα μπορούσε να συνδυαστεί με τα διαρθρωτικά ταμεία είναι ένας από τους τομείς στον οποίο βεβαίω προσπαθούμε να ε, διασφαλίσουμε σωστή σωστό συντονισμό πολιτικής. Σα ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα, κλείνουμε εδώ το σημείο αυτό. Ορίστε. Ορίστε. Ένα απάντηση, ε, μια απάντηση στην συνάδελφο Λέζινγκ. Διαβάζω τώρα το άρθρο 42, ε, παράγραφος 4 της συνθήκης τη μισή θα σας διαβάσω. Αποφάσεις, για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για, την, ε, ε, για τις αποστολές λέει ο ύπατος εκπρόσωπος θα μπορού, μπορεί σε, σε συνεργασία με την Κομισιόν να προτείνει τη χρήση εργαλείων μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέει μέσα στη συνθήκη είναι ένα εργαλείο της Ένωσης και μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα εργαλεία. Δεν έχει συμβεί αυτό κάτι στην πράξη, αλλά όταν έχουμε δορυφε, δορυφόρους, τον Κοπένικο, τον Γαλιλαίο, και υπάρξει ε, αποστολή στην Τουρκία για παράδειγμα για τη διάσωση των Κούρδων, θα έλεγα έτσι αυθόρμα, αυθόρμητα ότι αν έχουμε πάει εκεί για να σώσουμε ανθρώπους αλλά και για να προστατεύσουμε φυσικά και τους δικούς μας στρατιώτες ή ε, τους, ε, ε, ε, ανθρώπους μας που βοηθούν σε πολιτικά ζητήματα γιατί οι στρατιωτικοί δεν μπορούν πάντοτε να βοηθήσουν με τα υδροδοτικά ή τα ηλεκτρικά δίκτυα αν λοιπόν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο θα ήταν χαζό αυτό που βλέπουμε ήδη με τους δικούς μας δορυφόρες να μην το αξιοποιούμε για να πούμε ότι ναι εδώ υπάρχει ε, ένας κίνδυνος εδώ διότι το Ισλαμικό κράτος για παράδειγμα ε, χρησιμοποιεί ή στέλνει δυνάμεις στην τάδε περιοχή για παράδειγμα. Ναι, αυτό που λέω είναι ότι με τους δορυφόρους μπορούμε να έχουμε κάποιες πληροφορίες που μπορούν να μας βοηθήσουν. Με τους δορυφόρους μπορείτε να παρακολουθήσετε ε, πυρκαγιές σεισμούς, αλλά μπορείτε να παρακολουθήσετε και στρατιωτικές κινήσεις. Οπότε αν έχουμε κάνει την έρευνα η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί και να ωφελήσει στρατιωτικούς ή πολιτικούς σκοπούς, τότε για ποιο λόγο να μην τα αξιοποιήσουμε. Έχουμε το ίδιο εργαλείο τεχνολογικό με το οποίο μπορούμε να ε, επιδιώξουμε και πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους. Οπότε από αυτή την άποψη ναι, θεωρώ ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα να κλείσουμε τώρα αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης και να ευχαριστήσω τους δύο ομιλητές μας, τον ε, κύριο Ροζιέ και τον ε, κύριο Τοκάρσκι για την ε, πολύ περιεκτική παρουσίασή τους. Σίγουρα θα συνεχίσουμε την συζήτηση επί του θέματος αυτού στις επόμενες συνεδριάσεις μας την επόμενη χρονιά, κατά πάσα πιθανότητα. Ευχαριστώ λοιπόν. Οπότε τώρα αμέσως ε, περνάμε στο δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης μας που είναι οι εταιρικέ σχέσεις, η συμμετοχή γειτονικών χωρών στις ε, ενωσιακές αποστολές ε, στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Αλεσάνδρο Μαριάννη. Μαρίνη. Προϊστάμενο της διοικητικής μονάδας στην ε, Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της υπεύθυνη διοικητικής μονάδας που είναι ε, της που είναι υπεύθυνη μάλλον για την πολιτική κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και ο επόμενος ομιλητής είναι ο μη στρατιωτικό αντιπρόσωπος του Υπουργού Αμήνη τη Γεωργία, την κυρία Ταμάρ Κεκενάτζε και ο τρίτος ομιλητής είναι ο σύμβουλος στο πλαίσιο της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, ο κύριος Μπορίς Κρεμένσκι. Δίνω το λόγο πρώτα στον κύριο Μαρίνη για να μας κάνει μια εισαγωγή όσον αφορά τη συμμετοχή των ε, γειτονικών χωρών στις ε, αποστολές μας. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, εξοχότατοι εκπρόσωποι της Ουκρανίας και της Γεωργίας. Καταρχάς, θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε, καθώς και τους συναδέλφους σας, για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω σήμερα. Εννοείται ότι για μένα είναι μεγάλη τιμή Στην σημερινή μου παρουσίαση θα ήθελα να αρχίσω τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για στενή συνεργασία με εταίρους της στις αποστολές της ΚΠΑ. Είμαστε πεπισμένοι ότι η δυνατότητα, οι δικές μας δυνατότητες να συνεργαστούμε με άλλες εταιρικές χώρες είναι ουσιώδεις πολύ λίγα προβλήματα μπορούμε να λύσουμε μόνοι μας και αυτό ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για όλους τους άλλους. Πρέπει λοιπόν τους κοινού μας στόχους να τους προωθήσουμε μέσω πολυμερού συνεργασίας σε διεθνείς οργανισμούς και να συνάψουμε εταιρικέ σχέσεις με πολλούς εταίρους. Και γι' αυτό σήμερα χαίρομαι ιδιαίτερα που συζητούμε εδώ μαζί με εκπροσώπους της Ουκρανίας και της Γεωργίας. Η συνεργασία με τέρους είναι σημαντική από ενωσιακής απόψεως διότι αποτελεί τμήμα της συνολικής της προσέγγισης και διότι οι εταιρικέ σχέσεις μπορούν να βασιστούν στην τεχνογνωσία και τις δυνατότητες των εταίρων μας αλλά επίσης και να τους φέρουμε πιο κοντά μας. Είναι αυτή μια σημαντική πολιτική πτυχή λοιπόν που θα ήθελα να προσέξετε. Η Ένωση έχει αναπτύξει τέσσερα κλάστερ στην πολιτική της, της ΚΠΑ και θα ήθελα καταρχήν να τα ονοματίσω, να τα παριθμίσω ή να τα περιγράψω και μετά να περάσω στις λεπτομέρειες. Το πρώτο κλάστερ είναι εκείνο όπου υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί όπως το ΝΑΤΟ, ο ΙΕ κλπ. Το δεύτερο είναι εκείνο που θεωρούμε ως συμμετοχή σε δράσεις και αποστολές της ΚΠΑ. Τρίτο, πολύ συνδεδεμένο με το δεύτερο, είναι ο διάλογος για θέματα ασφάλειας και άμυνας και ο το τέταρτο είναι το capacity building που λέμε. Θα προσπαθήσω να σας τα περιγράψω ένα-ένα. Το πρώτο κλάστερ θα ήθελα επειδή θέλω να παραμείνω σύντομος να το αναφέρω σύντομα. Ας πούμε την εταιρική σχέση Ένωσης Ένωσης-ΟΙΕ είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για την Ένωση αλλά για όλους τους εταίρους μας. Για όλους. Οι εταίροι μας λοιπόν συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζουν παράλληλα πολύ καλά, ωφελούνται από αυτό που θεωρούμε πολύ μακροχρόνια και θετική συνεργασία για τη διαχείριση κρίσεων μεταξύ ΟΗΕ και Ένωσης. Ας πούμε. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ πριν από λίγους μόλις μήνες μετά από ε, μία από τις υψηλόβαθμες steering committees ήρθε να πληροφορηθεί στην Ένωση και όταν ρωτήσανε για την ποιότητα των σχέσεων με την Ένωση είπε ότι δεν είναι απλά μόνο σχέση, είναι τρόπος ζωής. Αυτό είναι σημαντικό γιατί σημαίνει ότι έχει συσσωρευτεί πολύ μεγάλη εμπειρία και στα θέατρα επιχειρήσεων όπως το Μαλί, τη Σομαλία, την Κεντρικοαφρικανική Δημοκρατία που συνοδεύεται και από υψηλού επίπεδου διάλογο και διαχείριση κρίσεων αλλά επίσης υψηλού επίπεδου συναντήσεις και επισκέψεις στη Νέα Υόρκη αλλά και την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Σύνοδο Ένωσης Αφρικής. Τώρα γιατί αναφέρομαι στις σχέσεις ΟΗΕ Ένωσης για τη διαχείριση κρίσεων διότι το σημαντικό μήνυμα που πάντοτε δίνουμε στους συνομιλητές μας είναι ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΟΗΕ και Ένωσης. Αντίθετα, υπάρχει διάλογος και επίτευξη συνεργασίας και συνέργειας για να αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε είδους κρίση. Θα επανέλθω σε αυτό αργότερα όταν θα μιλήσω για το παράδειγμα της παρέμβασης στην κεντροαφρικανική δημοκρατία που είναι και το θέατρο όπου και η Γεωργία αποφάσισε και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό να συμμετάσχει μαζί με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και όπως θα ξέρετε ε, ήταν πολύ σημαντική η συμβολή της Γεωργίας στο μπάνκι με πολλούς άντρες και γυναίκες. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο κλάστερ. Το δεύτερο, συμμετοχή σε αποστολές της ΚΠΑ και επιχειρήσεις, Φυσικά τα μέλη του ΝΑΤΟ και της Ένωσης είναι από τα πιο ενεργά στις δραστηριότητες και συνήθισαν και ορισμένες συμφωνίες πλαίσια που είναι εργαλεία για τη διευκόλυνση της συμμετοχής τρίτων χωρών σε επιχειρήσεις και αποστολές της ΚΠΑ υπό την καθοδήγηση της Ένωσης. 16 τέτοιες συμφωνίες υπάρχουν μέχρι σήμερα και περιλαμβάνουν την Αλβανία, τον Καναδά, τη Χιλή, την Κολομβία, τη Φιρόμ, τη Γεωργία, την Ισλανδία, το Μαυροβούνιο, τη Μολδαβία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ουρβηγία τη ε, Κορέα, την Νότια, Σερβία κλπ. Τουρκία κλπ. Ε, πέρα από αυτό το κατάλογο 16 χωρών, κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι πέρυσι είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε τέσσερις από αυτές τις συμφωνίες. Πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει μια τάση αυξανόμενου ενδιαφέροντος από άλλες τρίτες χώρες, εταιρικές χώρες, για τη σύναψη τέτοιου είδους συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γεωργία είναι μια από αυτές, διότι η συμφωνία με τη Γεωργία υπογράφτηκε πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, τον Νοέμβριο, στο, στη διάσκεψη του Βίλνιους. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν μερικές πληροφορίες για τη συμμετοχή εταιρικών χωρών, ατρίτων χωρών σε επιχειρήσεις και αποστολές της ΚΠΑ τους τελευταίους μήνες. Αυτά τα παραδείγματα τα διάλεξα για να, καταλα... για να γνωρίζετε κι εσείς να είναι πρόσφατα αλλά και για να φανεί ότι οι γειτονικέ χώρες είναι από τις πιο ενδιαφερόμενες και τις πιο διατεθειμένες να αναλάβουν ευθύνες από κοινού με την Ένωση για τη διαχείριση κρίσεων. Πρώτο παράδειγμα. Military operation in Central Africa. U4CAR στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Εδώ συμμετείχε και η Γεωργία με 154 ανθρώπους πράγμα που καθιστά τη Γεωργία τη δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη σε αυτή την αποστολή. Όταν λέω δεύτερη μεγαλύτερη, όχι με όρους μόνο τρίτων χωρών, αλλά με σε απόλυτους όρους. Η Γαλλία πρώτη και μετά η Γεωργία. Η uh, Η δημιουργία αυτή της Γεωργίας ήταν πλήρως λειτουργική και θα ήθελα να πω ότι σε κάθε ευκαιρία, με κάθε ευκαιρία την ευχαριστήσαμε πολλές φορές και φαντάζομαι ότι και εσείς συμφωνείτε ότι μπορούμε και σήμερα εκ νέου να την ευχαριστήσουμε. Τώρα, δύο άλλες έννοιες για αυτές τις επιχειρήσεις. Πριν από ένα χρόνο, εξετάζοντας την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, με τα λύπης μου λέω γιατί ήταν δύσκολα τα πράγματα, η κατάσταση θεωρούνταν προγενοκτονική κατάσταση. Αυτό βέβαια δεν έγινε η γενοκτονία, αλλά αν και είναι ακόμη νωρίς για να χαρούμε, εφόσον ακόμη βρίσκονται εκεί οι άντρες και οι γυναίκες της αποστολής και οι γεωργιανοί, θα έπρεπε να γνωρίζουμε ότι σε κάνα δύο χρόνια ακόμη θα μπορούμε να πούμε ότι η επιχείρηση αυτή Πράγματι άλλαξε τα πράγματα και σημαντικά, διότι η διάσωση ανθρώπινων ζωών νομίζω είναι κάτι το οποίο υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η επιχείρηση λοιπόν η New Car έδειξε ότι και η Τουρκία που συνέβαλε και αυτή με κάποια δύναμη έναν αξιωματικό στο Μπάγκι για τη δεύτερη κυρίως φάση. Και μετά η Σερβία που πρόσφατα έστειλε μια ιατρική ομάδα έξι ανθρώπων, έξι ατόμων. Άλλη επιχείρηση που θα ήθελα να αναφέρω, η Unifor Atalanta. Στην περίπτωση της Unifor Atalanta ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Ουκρανίας εδώ στα δεξιά μου, διότι η Ουκρανία στην αρχή του φετινού χρόνου από τις 3 Ιανουαρίου μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου συνέβαλε με μία ναυαρχίδα Σαβαντάτσνη λεγόταν με μία τορπιλάκα του έκανε πολύ καλή δουλειά και μάλιστα ο διοικητής του Γιουνάφορα Ταλάντα είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος και η συμβολή αυτή σημειώθηκε σε πολύ σημαντική χρονική στιγμή. Για γιατί το λέω αυτό, διότι σημειώθηκε στην αρχή αρχή της Προεδρίας της Ένωσης από την ομάδα επαφών για, κατά της πειρατείας στη θάλασσα. Για πρώτη φορά ανέλαβε τέτοιες ευθύνες η Ένωση. Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της είναι, θα είναι το 14 ο υπεύθυνο και η Προεδρία του οργανισμού αυτού από την Ένωση δείχνει ότι και η ίδια η επιχείρηση αλλά και ευρύτερα πολιτικά και διπλωματικά υπάρχει μεγάλη σημασία. Θα μπορούσα να σας πω πολλά για την ομάδα επαφών, αλλά όπως είπα γνωρίζω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεύτερη συμβολή στο UNAFOR από τη Νέα Ζηλανδία με ένα αεροπλάνο ναυτικής επιτήρησης και άλλες, από άλλες χώρες με ασυνοδευτικά πλοιάρια και με συμφωνίες μεταφοράς ή έκδοσης υπόπτων πειρατείας. Τώρα, τρίτο παράδειγμα, UTM Mali, η επιχείρηση UTM Mali. Εκεί υπάρχει μια κατάσταση όπου η Γεωργία σε λίγο θα στείλει δύο εμπειρογνώμονες έναν για ηλική υποστήριξη και τον άλλον σύμβουλο από την Άνοιξη. Υπάρχει και ένας εμπειρογνώμων από το, ναι, από το Μαυροβούνιο. Η Μολδαβία έστειλε κάποιον υπεύθυνο για ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ελβετία έναν ειδικό για μέσα ενημέρωσης και μόλις μάθαμε και δύο καινούργιες προσφορές. Δύο από τη Σερβία για μια ιατρική ομάδα τριών ατόμων και την Αλβανία με έξι. Και για να είμαστε πλήρεις ως προς τις συμμετοχές τρίτων χωρών σε επιχειρήσεις του τελευταίους 12 μήνες η Αυστραλία έστειλε έναν νομικό εμπειρογνώμονα στο Ιούκα Καπνέστορ Γενικά λοιπόν σήμερα έχουμε περίπου 560 ανθρώπους από τρίτες χώρες που συμμετέχουν σε αποστολές και επιχειρήσεις 8 περίπου δηλαδή της 100 της συνολικής δύναμης, των συνολικών δυνάμεων. Στην αρχή σας μίλησα για τρία κλάστερ. In mission and operation, but these... Αυτά πρέπει να τα συνδέσουμε και με τον διάλογο, με το κλάστερ για τον διάλογο. Διότι οι εταιρικέ σχέσεις είναι όλο και περισσότερο πολιτικά εργαλεία και γι' αυτό για μας όσο σημαντικές και να είναι οι συμβολές των τρίτων χωρών επίσης σημαντικές είναι, σημαντικός είναι και ο συνεχής διάλογος με τις χώρες αυτές. Σε αυτόν τον τομέα Θα ήθελα να, κάνω, να αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, στον διμερή διάλογο. Χώρες όπως η Γεωργία, η Ουκρανία, η Μολδαβία, ε, με, αυτές, αυτές χώρες έχουμε διμερή διάλογο. Και φέτος ξεκινήσαμε ε, διαβουλεύσεις, επίσημες διαβουλεύσεις ε, με την Μολδαβία. Με την Ουκρανία έχουμε ήδη εδώ και αρκετό καιρό αλλά ε, έπειτα από την ε, Σύνοδο Κορυφής της Βίλνιους τον Μάρτιο είχαμε αυτές τις διαβουλεύσεις οι, δια, οι διμερείς αυτές οι διαβουλεύσεις είναι πολύ σημαντικές γιατί μπορούμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή και να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε για παράδειγμα τη συμμετοχή χωρών σε επιχειρήσεις και αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητήματα που ενδιαφέρουν τους εταίρους μας, αλλά και πέραν αυτών έχουμε και ε, ένα φόρουμ πολυμερούς διαλόγου που είναι αυτό που κατά τη γνώμη μας συμπληρώνει τον διμερή διάλογο που έχουμε με χώρες όπως η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία. Και αυτός ο πολυμερής διάλογος ε, ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Είναι το πάνελ ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ε, της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος αυτού του πάνελ και πρέπει να σας πω να σας δώσω κάποιες πληροφορίες και κάποιες σκέψεις. Πρώτον, το πάνελ αυτό ξεκίνησε τις εργασίες του στο τέλος Σεπτεμβρίου πέρσι, οπότε και έγινε η πρώτη συνεδρίασή του. Αποφασίστηκε να συνεδριάζει, να συναντιάται αυτό το πάνελ κάθε έξι μήνες στην, ε, στις Βρυξέλλες. Γνώριζα βεβαίως εξ αρχής τι σημαίνει αυτό το διάστημα των έξι μηνών, αλλά δεν ε, περίμενα να υπάρχουν θέματα ε, έξι μήνες πριν τη συνεδρίαση. Όμως κάτι τέτοιο ε, συνέβη. Και αυτό οφείλεται και στο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από πλευράς των εταίρων. Έχουμε λοιπόν ε, φτάσει ήδη στην τρίτη συνεδρίασή μας. Πέρσι το Σεπτέμβριο ήταν η πρώτη, μετά η δεύτερη έγινε στο τέλος του Μαρτίου 2014 και η τρίτη συνεδρίαση έγινε τώρα στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2014. Και νομίζω ε, ότι γνωρίζω από τώρα που θα είμαι στα τέλη του Μαρτίου του 2015. Αυτό που είναι σημαντικό από ευρωπαϊκής ε, πλευράς είναι ότι πρόκειται για μια εργασία της Ένωσης διότι αυτές οι συναντήσεις δεν ε, αφορούν μόνο διάφορες επιρρησίες αφορούν και την ε, Κομισιόν, συμβάλλει και η Κομισιόν με την ΤΕΒΚΟ, έχει, υπάρχει μια αντιπροσωπεία του ε, Ευρωκοινοβουλίου στην ομάδα αυτή και υπάρχει και αντιπρόσωπος του Κολεγίου του Σώματος των Επιτρόπων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι η εκπαίδευση είναι σημαντικός πυλώνας ε, της στρατηγικής μας. Θα μπορούσα να σας δώσω πάρα πολλές λεπτομερείς πληροφορίες για το πώς ε, αυτό το φόρουμ λειτουργεί συγκεκριμένα. Μία σκέψη που θέλω όμως να σας πω είναι ότι πριν από ένα χρόνο όταν ξεκίνησε όλη αυτή η δουλειά μπόρεσα να ε, εντοπίσω ότι οι ομάδες είχαν εθνικό χαρακτήρα. Όταν λοιπόν είχα την δυνατότητα να γνωρίσω τους συναδέλφους από τις ε, χώρες εταίρους πήγαινα από τη μία ομάδα στην άλλη. Διότι οι άνθρωποι μιλούσαν με βάση την εθνικότητά τους. Αυτό δεν συμβαίνει πια. Σήμερα υπάρχει μια πραγματική ανάμιξη των, ε, των ε, συναδέλφων και αυτό είναι και ένα από τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι υπάρχει μια ανταλλαγή εμπειριών από όλες τις χώρες ε, προς όλες τις χώρες. Και με αυτό να ε, αναφερθώ και στο τελευταίο κλάστερ που ήθελα να αναφέρω αλλά για λόγους ε, πληρότητας της παρουσίασής μου θα πρέπει να σας πω επίσης ότι ε, υπάρχουν ότι τρεις ε, σύμβουλοι σε SSR έχουν αποσταλεί στην Μολδαβία που είναι και αυτό μια πολύ σημαντική ε, δράση. Το τέταρτο κλάστερ, εν πάση περιπτώσει, και με αυτό θα κλείσω και την παρέμβασή μου, είναι σχετικά με, ε, αφορά την ε, ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εταίρων. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους εταίρους μας με μονομένες χώρες και οργανισμούς ώστε να αναλαμβάνουν ευθύνες για την διαχείριση και την πρόληψη κρίσεων αυτόνομα. Αυτό είναι πολύ σημαντικός πυλώνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη υποστηρίζει περιφερειακές ή υποπεριφερειακές ε, οργανώσεις. Για παράδειγμα ε, υπάρχει η ε, Αφρικανική Αρχιτεκτονική Ασφάλειας, αλλά ασφαλεια αλλα εξαγάγει και πολύτιμα συμπεράσματα από τη Σομαλία και το Μάλι. Η εκπαίδευση λοιπόν ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο για την ε, κατάρτιση αυτής της αρχιτεκτονικής. Η εκπαίδευση λοιπόν των ε, δυνάμεων ασφαλείας είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ήθελα να πω ότι οι προσπάθειές μας θα πρέπει να κατατείνουν στην αξιοποίηση διαφόρων εργαλείων που θα συνδυάζουν την ασφάλεια και την ε, ανάπτυξη. Φυσικά πρέπει να τηρούμε 100% τους κανονισμούς μας, αλλά όλο και περισσότερο τονίζεται στη διεθνή κοινότητα αυτή η σχέση μεταξύ ανάπτυξης και ασφάλειας. Δεν υπάρχει δηλαδή ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη, αλλά δεν υπάρχει και ανάπτυξη αν δεν υπάρχει ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πλήρη παρουσίαση. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από την κυρία Ταμάρκα Κνάτσα να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όπως και ο κύριος Μαριάννη διότι μαζί να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ε, τα θέματα της ε, συνεργασίας σε θέματα άμυνας. Ε, όπως πολύ εξαιρετικά παρουσίασε ο κύριος Μαριάννη τις διάφορες μορφές συνεργασίας μας, η φετινή χρονιά ήταν πολύ σημαντική διότι υπήρξε η υπογραφή της συμφωνίας που επέτρεψε στην Γεωργία να συνεισφέρει περισσότερο στην ασφάλεια Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας και τη, την ασφάλεια πέρα από τα σύνορα. Ε, μας δόθηκε η δυνατότητα επίσης στη διάρκεια του έτους να συμμετάσχουμε σε, ε, στις δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, αποστολή στην Κεντρική Αφρική. Ε, η Γεωργία είχε δύο δημιουργίες ήδη στο Αφγανιστάν και υπήρξε και μία ακόμα μονάδα που ήταν για τις ομάδες ε, δράσης του ΝΑΤΟ. Και σε γενικές γραμμές η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προσπάθειές μας για την ε, συνέχεια ε, της ε, διεθνούς ασφάλειας ήταν αποφασιστική σημασίας και ήταν θετικά τα θέματα της συμμετοχή μας. Θα ήθελα να τονίσω ότι όταν το Κοινοβούλιο συζητούσε το κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή στην αποστολή μη, ελήφθηκε ομόφωνα απάντηση από ε, τη Γεωργία και η πλειονότητα του πληθυσμού στη Γεωργία υποστήριζε αυτήν την ε, πρωτοβουλία. Ταυτόχρονα μας είχε χαροποιήσει και ιδιαίτερα το γεγονός ότι μπορέσαμε λίγο να ξεπληρώσουμε τη στήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι από το 2008 λαμβάναμε ε, υποστήριξη μέσω της ε, ε, συμφωνίας για την ε, ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα εδώ επί ευκαιρία να σας ευχαριστήσω διότι η ομάδα παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μόνη διεθνής οργάνωση που είναι παρούσα στη κατεχόμενα εδάφη. Ε, το Κοινοβούλιο με τους βουλευτές αποφάσισαν λοιπόν κατά πόσον θα πρέπει να συμμετέχουν στην αποστολή για την Κεντρική Αφρική και αυτή η δυνατότητα ε, Μα δόθηκε και χαίρομαι ιδιαίτερα και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση γιατί τα πάντα εξελίχθηκαν ομαλά και χωρί την υποστήριξή του δεν θα μπορούσαμε να είχαμε ε, τόσο καλά αποτελέσματα. Ήταν η πρώτη φορά για μα που χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία, αν μου επιτρέπετε. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και ε, όταν θα ολοκληρωθεί η αποστολή θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τι διδάγματα αντλήθηκαν με τους εταίρους μας και όπως είπε και ο κύριος Μαρίαν είμαστε έτοιμοι να στείλουμε και δύο ε, υπαλλήλους ε, στην Ευρωπαϊκή ε, αποστολή εκπαίδευσης ε, στο Μάλι. Ένας θα φύγει φέτος και ένας δεύτερο θα πάει του χρόνου. Ο κύριος Μαριάννη ουσιαστικά με πρόλαβε σε όλα όσα ήθελα να πω, επομένως εγώ δεν θα πω πάρα πολλά στην παρουσίασή μου και απλώς ε, θα σας πω τι αίσθηση έχουμε εμείς για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα άμυνας, διότι αυτό είναι συμπληρωματικό της όλης συνεργασίας Γεωργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Προσβλέπουμε λοιπόν στις διμερείς συζητήσεις με τους εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής ε, Δράσης αυτό το μήνα στη Γεωργία. Ε, διερευνούμε πολύ, περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας, όχι μόνο σε θέματα συμμετοχής επιχειρήσει επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, αλλά και σε άλλους τομείς που θα μπορούσαν να είναι προς όφελος και των ε, κρατών μελών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων μας να τονίσω ε, τη σημασία του πάνελ κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Αυτό άλλωστε τονίστηκε. Αυτό το πάνελ μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τους εταίρους και γειτονές μας και φυσικά να μάθουμε και εμείς από αυτούς έχοντας κατά νου φυσικά και τι ε, θέματα ασφαλείας υπάρχουν στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυνατότητα. Θα είμαι πολύ σύντομη, είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Κραμίτσκι. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, Uh, e είμαι ο ταξίαρχος Κρεμέτσκι και θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ σύντομος. Από την ανεξαρτησία της η Ουκρανία θεωρεί τη συμμετοχή της στη διαχείριση διεθνών κρίσεων ως συμβολή της προς την εθνική της ασφάλεια. Και συμμετέχουμε ενεργά σε διαχείριση κρίσεων παγκοσμίως προσπάθειες του ΟΗΕ στην Αφρική, συμμετέσχομαι σε όλες τις αποστολές, πρόσφατες αποστολές του ΝΑΤΟ και το 2005 υπογράψαμε μία συμφωνία με την Ένωση, συμφωνία πλαίσιο για την ασφάλεια που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ανταλλαγές απόψεων και πληροφοριών ε, αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Από τότε η Ουκρανία προσπαθεί να είναι δραστήρια σε αποστολές της Ευρωπαϊκής ε, ΚΠΑ όπως η αποστολή Γιούπολ στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη όπου στείλαμε 5 με 12 αστυνομικούς μέχρι το τέλος της αποστολής της επιχείρησης. Το 2008 εκλήθη η Ουκρανία να συμμετάσχει στις προσπάθειες της Ένωσης για την καπολέμηση της πυραμίας και εστάλθηκε ένας Ουκρανός αξιωματούχος. Συνεργαστήκαμε με αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό για την προστασία πλοίων στην επιχείρηση Αταλάντα. Δυστυχώς η συμμετοχή τελικά ακυρώθηκε για λόγω κάτι νομικών προβλημάτων. Δεν μπορέσαμε να στείλουμε το αεροπλάνο που αναφέρθηκε πριν. Αλλά αποφάσισαν οι Ουκρανικές αρχές να στείλουν μια φρεγάτα παρόλα αυτά. Για έξι μήνες. Και τους πρώτους τρεις μήνες στην επιχείρηση του ΝΑΤΟ Ocean Shield και δύο άλλους μήνες στην Αταλάντα. Για την Ουκρανία αυτό ήταν μια πολύ χρήσιμη εμπειρία. Η φρεγάτα μας ε, έκανε ό,τι τη ζητήθηκε όπως προβλεπόταν από τους κανόνες της επιχείρησης. Επιτηρούσαμε την περιοχή και προστατεύαμε εμπορικά πλοία παρεμποδίζοντας τη δράση των πειρατών. Η Ουκρανική λοιπόν αυτή δύναμη που συμπεριλάμβανε και ένα ελικόπτερο, το, το, το προσωπικό της φρεγάτας και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό ανήλθε σε 250 άτομα μαζί με το ελικόπτερο. Καλύψαμε 10.000 χιλιόμετρα και 45 ημέρες επιχειρήσεων θα έπρεπε να σας πω ότι η Ουκρανία είναι ο μεγαλύτερος αναχώρα συνεισφέρον και οικονομικά σε επιχειρήσεις από, σε τέτοιες επιχειρήσεις από την ανεξαρτησία μας και μετά. Αν θεωρήσουμε ότι η Αταλάντα είναι επιτυχία τότε και η Ουκρανία συνέφερε στην επιτυχία αυτή. Ακόμη αναλύουμε τα μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε από αυτή την επιχείρηση, αλλά ήδη μπορούμε να πούμε ότι καταφέραμε να πετύχουμε στενή συνεργασία με όλους τους οργανισμούς της Ένωσης και της Στρατιωτικής Επιτροπής καθώς και όλους τους υπόλοιπους θεσμούς και όργανα. Για να συντομεύω θα έλεγα ότι η Ουκρανία είναι δεσμευμένη να συμμετάσχει και στο μέλλον σε τέτοιες επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ένωσης. Η Συμφωνία Σύνδεσης με την Ένωση που πρόσφατα εγκρίθηκε και από το Ευρωκοινοβούλιο και από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο μας δίνει περισσότερα εργαλεία και μέσα για τέτοιου είδους συμμετοχές και αν υπάρξουν ερωτήσεις με τα χαρά να σας απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κρεμενέτσκι. Πρωτού δώσω το λόγο για να ξεκινήσει η συζήτηση θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, η Γραμματεία και ο Πρόεδρος έχουν πρόθεση να προσκαλέσουν και άλλους ε, ε, εταίρους. Πρώτα και κύρια τη Μολδαβία, για να συζητήσουμε τις προσπάθειες στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Και δεύτερον, ότι και οι δύο χώρες, η Ουκρανία, αλλά και νωρίτερα η Γεωργία, έχουν συμβάλει πολύ σημαντικά στις προσπάθειές μας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, παρά την πολύ δύσκολη ε, κατάσταση όσον αφορά την ε, ασφάλειά τους. Στην Ουκρανία υπήρξε εξωτερική επέμβαση, στρατιωτική. Παρόλα αυτά η Ουκρανία παραμένει δεσμευμένη και το ίδιο συμβαίνει και στην ε, περίπτωση της Γεωργίας, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η απειλή κατά των συνόρων και της εδαφικής ακαιρεότητας της χώρας. Παρόλα αυτά η Γεωργία εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά, ενεργότατα στις ε, προσπάθειές μας. Και τώρα μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. Κύριε Γέλλερ, συντονιστές από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομος θα είμαι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας για αυτές τις πολύ ε, ολοκληρωμένες παρουσιάσεις και εγώ μέχρι τώρα δεν γνώριζα σε ποια έκταση συνεργαζόμαστε με τις τρίτες χώρες, σε ποιο βαθμό και νομίζω ότι ο κύριος Μαριάννη ε, περιμένετε ακόμα για τη διερμηνία την ψάχνετε α, μόλις τη βρήκατε, ωραία κανάλι 4 για εσάς κύριε Μαριάννη. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ λοιπόν για, τις, ε, για τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε και νομίζω ότι ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το εργαλείο αυτό ως αυτό που είναι στην πραγματικότητα και το είπατε. Πρόκειται για συμμετοχή και η συμμετοχή είναι πολιτικό εργαλείο. Και στόχος μας είναι επίσης βεβαίως ο μόνιμος διάλογος και αυτές είναι οι δύο παράμετροι για να μπορέσουμε και εμείς να δείξουμε ότι με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας μας ασκούμε μία πολιτική που έχει θετικές απο, επιπτώσεις και αποδοχή και σε άλλες χώρες και ταυτόχρονα προβαίνουμε και σε διάλογο, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα, ειδικά σε περιόδους κρίσης, να κατανοούμε τους εταίρους μας. Και ελπίζω στο πλαίσιο αυτό ότι οι προσπάθειες αυτές θα συνεχιστούν και στο μέλλον και μάλιστα θα συμπεριλάβουν και άλλους εταίρους. Θα μπορούσα για παράδειγμα να φανταστώ στην στη νότια πλευρά της Μεσογείου την Τινησία που είναι μια χώρα που είναι ένας παράγοντας σταθερότητας στην ε, περιοχή και να, θέσω και ένα ερώτημα. Έχετε σκεφτεί μια πιθανή συνεργασία στον τομέα αυτό με την, ε, την Ισία. Ευχαριστώ. Η κυρία Λέζιν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις αυτές. η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να συμπεριλάβει σε αυτές τις προσπάθειες, σε αυτές τις επιχειρήσεις όσο και περισσότερο. Ο κύριος ε, ο προλαλήσαντας ε, μάλιστα μας παρέπεμψε και σε πιθανό, πιθανές διευρύνσεις ε, αυτών των προσπαθειών με άλλα κράτη. Αυτή τη στιγμή, ε, από ό,τι καταλαβαίνω, ε, υπάρχουν 45 κράτη που έχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμμετάσχει σε επιχειρήσεις και αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκουσα τις παρουσιάσεις για τη Γεωργία και την Ουκρανία και διάβασα και τα έγγραφα που μας στείλατε συνοδευτικά προς αυτήν την συνεδρίαση. Υπάρχει και μάλιστα ε, ένα έγγραφο του Ινστιτούτου Έρευνας ε, για την συμπερίληψη νέων τρίτων χωρών. Και εδώ τα πράγματα μάλλον περιγράφονται διαφορετικά. Λέγεται, αναφέρεται εδώ ότι όταν συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλές ε, χώρες τότε τα ωφέλη είναι πάρα πολύ μικρά και ότι είναι πολύ δύσκολο να ε, να αξιοποιηθούν τα ωφέλη αυτά και ότι ταυτόχρονα είναι και πολύ, έξοδα τα, ε, πολύ ε, υψηλά τα έξοδα. σε αυτό το έγγραφο, για παράδειγμα, χαρακτηρίζονται και ως δευτεροκλασάτες ε, κάποιες χώρες που μάλιστα δεν έχουν, την, δεν έχουν λόγο στη διαμόρφωση των επιχειρήσεων και των αποστολών. Έτσι λέει το έγγραφο. Οπότε ξαναθέτω εγώ το ερώτημα. Ποια είναι τελικά τα ωφέλη από αυτήν την ενσωμάτωση, την συμπερίληψη νέων χωρών στις επιχειρήσεις και στις αποστολές μας. Ο κύριος Μαριάννη και οι άλλοι ομιλητές είπαν ότι είναι πολιτικοί οι λόγοι, ε, ότι ενισχύονται οι εταιρικέ μας σχέσεις. Εγώ θα ήθελα να σας πω τη δική μου άποψη και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του κυρίου Μαριάννη επί της δικής μου άποψης. Μήπως υπό ορισμένε προϋποθέσεις θα ε, μπορούσαμε να μιλήσουμε και για μια ε, σύγκληση των οπλικών συστημάτων. Μήπως τελικά αυτή η συνεργασία στο πλαίσιο των αποστολών συμβάλλει στην σύγκληση των οπλικών συστημάτων, μήπως δε στόχος ε, τελικά είναι να ισχυθούν οι πωλήσει ε, οπλικών συστημάτων ε, Ευρωπαίων κατασκευαστών σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Thank you, Mr. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στέτινα. Ευχαριστώ πολύ. έχω μια ερώτηση για όλο το πάνελ, αλλά κυρίως για τον κύριο Κρεμιέσκη. Την περασμένη εβδομάδα ο πρώην Πρωθυπουργό Κάρλ Σβάρτ στην ε, Τσεχική Δημοκρατία, που είναι και επικεφαλή του κόμματο το οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είπε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την Ουκρανία με πολύ περισσότερα και να μην επιβάλλουμε απλώ κυρώσει. Ο κύριος Σάντσπερκ ζήτησε η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει και όπλα και θα ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας για την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή μου είναι αν Πραγματικά πρόκειται απλώς ε, για μία ποσοτική συγκέντρωση και όχι μία ποιοτική αξιολόγηση αυτά τα οποία συζητούμε. Και τι εξηγώ, εξηγώ τι εννοώ. Ε, μου φαίνεται ότι μάλλον είναι ε, ακαδημαϊκή προσέγγιση αυτό που κάνουμε και όχι πρακτική λύση επιτόπου. Και θα σας μιλήσω για δύο θέματα. Ε, η κεντροαφρικανική δημοκρατία Καταλαβαίνω πολύ καλά τι κάνει η Γεωργία και το κάνει καλά, αλλά είπατε εσείς ότι απεφεύχθηκε η γενοκτονία. Η Κεντρική Αφρική δεν είναι μόνο η πρωτεύουσα. Υπάρχει η Νταρούγκα, το Μπαγκασού, πρόκειται για περιοχές τις οποίες δεν έγινε τίποτα, δεν είδατε τίποτα και εκεί ε, σας ε, ε, ανακοινώνω ότι υπήρξε γενοκτονία, έγινε εθνοκάθαρση. Και νομίζω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο ευχαριστημένοι με την ύπαρξή μας, διότι κάναμε κάτι σημαντικό, δηλαδή το Μπαγκί να γίνει ε, μια περιοχή στην οποία υπάρχει απλώς εθνική καταστροφή. Έγινε μόνο στο Μπαγκί όμως αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Μου φαίνεται εξαιρετικό ε, το να ε, περιλαμβάνουμε διάφορες ε, μονάδες, μίνι μονάδες, ε, για να μας μιλήσουν για προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ε, ε, δικαιωμάτων των γυναικών στην δημοκρατία του Μάλι. Αλλά στο ΣΑΙΔ, στο Κιντάλ δεν είναι θέμα ισότητας φύλων, ούτε θέμα νομικό, ούτε τίθεται θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταφυσικών τα οποία καταλήγουν στην πόρτα του κέντρου εκπαίδευσης στον Παμάκο. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και επειδή ακριβώς ε, στις περιοχές αυτούς ε, φτάνουν και μονάδες εκπαίδευσης, εμένα πραγματικά με αφήνει άναυδο, απόλυτα άναυδο το γεγονός ότι εμείς κάνουμε και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλό μία εκπαίδευση απλώς και μόνο διαδικαστική για ε, παραστρατιωτικές ε, δράσεις στην περίπτωση του Μάλι και όταν έρχονται αντιπέτωποι με την πραγματική στρατιωτική παρέμβαση δηλαδή την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας στην περιοχή του Κιτά, του Καταοτενή, σε όλη την ευρύτερη περιοχή πραγματικά ε, χάνονται στα εξών συνετέθησαν πάρα πολύ εύκολα, διότι δεν, ξέρουν, ε, δεν έχουν καμία εκπαίδευση. Υπάρχει, ξέρετε, ποια είναι η καλύτερη στρατιωτική ομάδα σε επιχειρήσεις στη Σαχάρα και με εκπλήσει το γεγονός ότι υπάρχουν στρατιωτικές μονάδες που δεν ξέρουν ε, καθόλου τι σημαίνει ε, μάχη στην έρημο της Σαχάρας και γίνονται με μονάδες που δεν έχουν δει ούτε άμμο, ούτε ξέρουν τι σημαίνει να δίνει κάποιος μονά, ε, μάχη στην άμμο με μικρές ε, μονάδες που πραγματικά δεν έχουν καθόλου δυνατότητες επιμελητίας. Και αυτό κάνει ο γαλλικός στρατός αλλά με βαριά επιμελητία. Και πραγματικά σας ρωτώ, Συζητάμε δόλο φιλοσοφικά και μεταφυσικά ζητήματα. Γιατί δεν σκεφτήκατε να συμπεριλάβετε το μόνο στρατό που ξέρει τι να κάνει στην έρημο, που είναι αυτό που έλυσε και το πρόβλημα στο Μάλι, που είναι ο στρατό του Τσάντ. Θα ήθελα να κάνω ένα θερμό ε, χαιρετισμό σε όλους τους προσκεκλημένους μας για αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα ζητώματα και θα ήθελα να πω ότι η Ουκρανία και η Γεωργία είναι δύο παραδείγματα, σαφέστατα παραδείγματα, ε, χωρών που βιώνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι ένοπλες δυνάμεις και οι πολιτικές δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ε, υπερασπιστούν την ε, κυριαρχία τους. Και αυτά τα παραδείγματα μας δείχνουν ενθαρρυντικά ότι οι δύο αυτές χώρες μπορούν και συμμετέχουν και σε πολύ δύσκολες αποστολές. Εκ να σας πω ότι ήταν εξαιρετική η συνεργασία με τους συναδέλφους από την Ουκρανία και από τη Γεωργία στο Ιράκ και πιο συγκεκριμένα η ταξιδιαρχία της Ουκρανίας και υπήρχαν και εξαιρετικές εμπειρίες με τους συναδέλφους από τη Γεωργία. Mm. Και δεν είναι αλήθεια ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν τη διάθεση, τη δύναμη ε, και τους στρατιώτες που μπορούν να δράσουν πολύ αποτελεσματικά και μάλιστα και σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Αλλά θα ήθελα λίγο να αναστρέψω την κατάσταση. Η δράση των χωρών αυτών είναι πάρα πολύ θετική, αλλά θα ήθελα να θέσω και δύο ερωτήσεις για να ταράξω και λίγο τα νερά. Όλες αυτές οι αποστολές είναι πάρα πολύ σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την κάθε χώρα φυσικά, αλλά αυτές οι αποστολές είναι πάρα πολύ σημαντικές και για χώρες που στέλνουν τους στρατιώτες τους. Επομένως, θα ήθελα να θέσω την εξή ερώτηση. Αυτή η εμπειρία της συμμετοχής στις ε, διεθνείς αποστολές χρησιμοποιείται προκειμένου να ενισχυθούν ε, οι ένοπλες δυνάμεις της κάθε χώρας και ε, δεύτερη ερώτηση, η οποία έχει σχέση και με την πρώτη. Αυτή η αποστολή εκπαιδεύει στρατιώτες αλλά και διοικητές. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον λοιπόν οι Ουκρανοί και οι Γεωργιανοί στρατιώτες που συμμετείχαν σε αυτές τις αποστολές έχουν ε, στη συνέχεια και προαγωγές πιο γρήγορα στην, ε, σε ενοπλές Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους ομιλητές μας, να ξεκινήσω με τον κύριο Μαρίνη, να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις και μετά θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Κεκνάτσε και στον ε, υποστράτηγο. Thank you very much. First of all, Ευχαριστώ πολύ για την πρώτη ερώτηση του κύριου Γκάλερ. Ναι, ο διάλογος είναι βασικό στοιχείο, όπως ακριβώς ε, τονίσατε και εσείς, και ιδιαίτερα αυτού του είδους η συνεργασία ναι βεβαίως εξετάζουμε τους γείτονές μας και όχι μόνο τους, ε, ε τις χώρες της Ανατολικής Συνεργασίας οπότε για να σας ενημερώσω ενεργούμε στη βάση εντολής του Συμβουλίου και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαβουλεύσεις, σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο. Αυτά για να απαντήσω στο ερώτημα σας και στην παρατήρησή σας ότι θα πρέπει να εξετάζουμε τους ε, γείτονές μας στην ε, Μεσόγειο με την ίδια ε, θέρμη όπως κοιτάζουμε τους ε, ανατολικούς μας εταίρους. Και εγώ θα ε, έθετα και τις, τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Το δεύτερο ερώτημα αφορούσε το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Μελετών για την Ασφάλεια. Γνωρίζετε ότι το Ινστιτούτο αυτό είναι πλήρως ανεξάρτητο Σε κάποια από αυτά τα στοιχεία του άρθρου ε, συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει μια δημοσιογραφική επιθυμία και ενδεχομένως να χρησιμοποιείται και πολύ ε, έντονη διατύπωση. Το κόστος, το ότι το κόστος είναι υψηλό είναι μάλλον μια δήλωση που με εκπλήσει. Διότι πρέπει να σας ενημερώσω ότι κάθε ε, κάθε χώρα συμβάλλει ε, οικονομικά στις αποστολές, στις συνεργασίες αυτές. Γνωρίζετε ότι σε κάθε ε, στρατιωτική επιχείρηση ε, το κόστος ε, βαρύνει την αρχή που αποστέλει δεν πρόκειται δηλαδή για ένα κόστος που ε, αφορά αποκλειστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, όταν ευχαριστούμε τους εταίρους μας για τη συμμετοχή τους, ακριβώς αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει και μια οικονομική προσπάθεια από την δική τους ε, πλευρά. Αναφερθήκατε σε δευτεροκλασσάτους παίκτες. Νομίζω ότι πρόκειται για μια πολύ ε, απαρχαιωμένη αντίληψη για τη συμμετοχή των ε, τρίτων χωρών. Έχουμε κάνει πολλά για να ε, μην υπάρχει μια τέτοια συμπεριφορά. Για παράδειγμα, πληροφορία α όταν θέλουμε να συνάψουμε μια εταιρική σχέση βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο διάλογος γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και έγκαιρα τις ε, πληροφορίες. Αυτό που λέει το άρθρο είναι ότι προσπαθούμε να ε, γεμίσουμε κενά. Αλλά αυτό δεν ισχύει σήμερα. Όταν προετοιμάζουμε επιχειρήσεις, βρισκόμαστε σε διαβουλεύσεις με τους εταίρους μας και ξέρουμε εκ των προτέρων αν θέλουν να συμμετάσχουν στην επιχείρηση ή όχι. Και εκείνοι μπορούν στη συνέχεια να μας εξηγήσουν ότι... Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα γίνονται πάρα πολλές ε, συναντήσεις εκ των προτέρων, αλλά δεν μπορούν να, να είναι να καλύπτουν και την τελευταία λεπτομέρεια, γιατί πολλές φορές προκύπτουν ζητήματα που πρέπει να λαμβάνει κανείς αποφάσεις ad hoc. Τώρα, ποια είναι τα ο, ο, ωφέλη. Θα έλεγα τρία. Νομιμοποίηση, διότι είναι πάντοτε καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει και άλλες χώρες που συμμετέχουν στις δικές της ε, δράσεις και δημιουργούμε συνθήκες όπου οι εταίροι μας είναι πολύ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το άλλο στοιχείο είναι ο διάλογος διότι όπως είπα η συμμετοχή από μόνη της είναι μεν σημαντική αλλά δεν είναι ο τελικός μας στόχος. Δεν είναι ο τελικός στόχος. Ο τελικός μας στόχος είναι να υπάρχει ένας διάλογος μέσα από τον οποίο θα μπορούμε να προσδιορίζουμε από κοινού λύσεις και να ε, καταφέρνουμε να επιλύουμε διάφορες ε, κρίσεις με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Δεν υπάρχει η πρόθεση να πουλήσουμε οπλικά συστήματα, δεν υπάρχει εμπορική διάσταση καθόλου και πρέπει να σας, να σας ομολογήσω ότι εγώ προσωπικά δεν, δεν μου έχει τύχει ποτέ να τεθεί τέτοιο ζήτημα. Το τρίτο ερώτημα, αν κατάλαβα σωστά, αφορούσε τον Ουκρανό συνάδελφο. Συμφωνώ απόλυτα πάντως με τον Ισπανό Ευρωβουλευτή Το είπα αλλά ίσως δεν κατάφερα να το διευκρινίσω επαρκώς. Ήθελα να πω ότι σε λίγα χρόνια ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να δούμε ότι έχουμε επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα και ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Είναι γεγονός ότι πρόκειται για μια επιχείρηση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης Κεντρικής Αφρικής, ε, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και του ΟΗΕ συνέβαλε για μια μεταβατική περίοδο ώστε ο ΟΗΕ να μπορέσει να αναπτύξει τη δική του αποστολή η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από τα μέσα του Σεπτεμβρίου και ακριβώς επειδή είναι πολύ μεγαλύτερη η αποστολή του ΟΗΕ ως προς το προσωπικό μπορεί βεβαίως να καλύψει πολύ περισσότερα ζητήματα. Συγγνώμη ε, αν, έδωσα την εντύπωση ότι ε, επιχείρησα να υπερτονίσω τα θετικά αποτελέσματα. Πιστεύω ωστόσο ότι υπάρχει και μια κάποια συλλογική ε, ευθύνη να παρουσιάζουμε με δίκαιο τρόπο τα αποτελέσματα που αποφέρει η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν υπάρχουν θετικά αποτελέσματα δεν θα πρέπει να διστάζουμε να τα λέμε. Το δεύτερο θέμα που θέσατε, η απάντηση είναι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει τον μέγιστο δυνατό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει ούτε αλλά, ούτε αν, ούτε οτιδήποτε, οποιοδήποτε άλλος σύνδεσμος. Αναφερθήκατε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των αξιωματούχων της δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ τα μάτια της μπροστά σε καταστάσεις που χρειάζονται την προσοχή μας και μάλιστα την πολύ σοβαρή προσοχή μας. Από αυτή την άποψη, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η εκπαίδευση στρατιωτικών μονάδων από την UTM στο Μάλι είναι εξαιρετική. Κανείς τους, εξ όσων γνωρίζω, δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να τους θέσουν σε κίνδυνο όπως αυτές οι μονάδες εκπαίδευσης που αναφέρατε. Αλλά θέλω επίσης να πω ε, ότι η προσοχή που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ανθρώπινα δικαιώματα και, και στην ισότητα των φύλων σε κάθε αποστολή έχουμε ένα άτομο υπεύθυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων και όποτε τίθεται, ανακύπτει ανάγκη, βρισκόμαστε σε συνεργασία στενή με αυτόν τον συνάδελφο. Δίνουμε λοιπόν τη μέγιστη προσοχή, διότι αυτές είναι οι θεμελιώδεις αρχές ε, για τη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών. The last, Για τα τελευταία δύο ερωτήματα... Νομίζω ότι θα είναι καλύτερα να απαντήσουν ε, ο συνάδελφος από την Ουκρανία και ο συνάδελφος από την Γεωργία. Ο κύριος παρακαλώ. Η κυρία. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας σε αυτά τα θέματα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, να απαντήσω σύντομα σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούσαν τη Γεωργία και τη συνεργασία μας με την Ένωση. Το θέμα της ποιότητας έναντι της ποσότητας είναι σημαντικό θέμα και εμείς προσέχουμε να επιλέγουμε όποιον θα στείλουμε σε διεθνείς επιχειρήσεις με μεγάλη προσοχή. Η Γεωργία συμμετέχει από το 1999 σε τις επιχειρήσεις του Κοσυφοπέδιο, Ιράκ και τελευταία και στο Αφγανιστάν. Στο Αφγανιστάν έχουμε στείλει πάνω από 12.000 ανθρώπους με μεγάλη στρατιωτική εμπειρία και η μονάδα που στείλαμε στην Κεντρική Αφρική Είχε επίσης εμπειρία από το Αφγανιστάν. Γι' αυτό θεωρούμε ότι ωφελήσαμε την αποστολή και την επιχείρηση. Και όσοι πήγαν εκεί μάθανε πολλά και από τους Γεωργιανούς. Τον περασμένο Αύγουστο ο υπουργό Αμήνης μας πήγε επί τόπου και ως προς τα μαθήματα που πήραμε και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον για την εκπαίδευση τέτοιων στρατιωτών. Θα τα πάρουμε όλα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Ήδη αυτό έγινε για την αποστολή στην Κεντρική Αφρική, αν και δεν τελείωσε ακόμα. Και θα γίνει μια τελευταία αποτίμηση και όταν τελειώσει η αποστολή επιχείρηση το Δεκέμβριο ως προς το κόστος και τους πόρους πράγματι αλήθεια είναι ότι είναι ακριβό υψηλό το κόστος. Προσπαθούμε όμως να διατηρήσουμε ορισμένα πρότυπα σταθερά. Όταν αναλαμβάνουμε πρόσθετο δημοσιονομικό βάρος, όπως όταν στείλαμε δύο δημιουργίες στο Αφγανιστάν και αλλού θεωρούσαμε ότι αυτό ήταν για μας μια ευκαιρία να προωθήσουμε τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συμβάλλουμε και εμείς και χαρήκαμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Άλλο ερώτημα ήταν τα battle groups. Εδώ θα θέλαμε να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θα είναι ένα από τα θέματα των συζητήσεών μας το Νοέμβριο. Τέλος, κάτι που δεν το είχατε απευθύνει σε μένα, για την υποστήριξη η Ουκρανία δεν θέλω να πω τι είδους υποστήριξη πρέπει να χορηγήσει γιατί τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα το καθορίσουν αυτό για την Γεωργία όμως εμείς είχαμε πολύ στενή συνεργασία με την Ουκρανία και προσπαθήσαμε να τους υποστηρίξουμε όσο περισσότερο μπορέσαμε σε πολλούς τομείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Ο κύριος ε, Κρανιέτσκι. Α, ένα πολύ σύντομο διαδικαστικό. Ναι, Πρόκειται για διαδικαστικό ζήτημα, διότι δεν μου απαντήσατε. Εγώ σας ρώτησα, κυρία Μαριάννη, δεν μου απαντήσατε. Μπορεί να μην ε, εκφράστηκα σωστά. Εγώ αναφέρθηκα σε πρακτικές λύσεις. Εγώ σας είπα ότι έξω από την πόρτα του στρατοπέδου στο οποίο εκπαιδεύονται οι δημιουργίες του Μάλι ε, τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητα των φύλων είναι θέματα τα οποία δεν είναι και τόσο σημαντικά και οι άνθρωποι που εκπαιδεύουμε δεν ε, κάνουν επιχειρήσεις επιτόπου και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, το γνωρίζουμε και αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται αντιπέτωποι με τρομοκράτες και με Ισλαμιστές τρομοκράτες. Και ερώτησή μου είναι εάν πέρα από ακαδημαϊκά στρατιωτικά ζητήματα να ζητούμε και μια αποτελεσματική, πραγματική ε, συνεργασία γιατί για να δώσει κάποιος μάχη στην έρημο χρειάζεται εμπειρία και αν κάποιος έχει ε, ε, να δώσει μάχη με ε, ε, ε, με άμμο, με νερό το οποίο προέρχεται από πηγάδια και δεν προέρχεται από πουθενά αλλού. Γιατί δεν δίνουμε στρατιωτικές δυνατότητες ε, και έχουμε στρατό ο οποίος δεν είναι έμπειρος, με εξαίρεση το γαλλικό στρατό και δεν ξέρει να δίνει μάχες στην έρημο και γιατί δεν χρησιμοποιούμε το στρατό του Τσάντ που είναι ο στρατός ο οποίος έβγαλε τα κάστανα στη φωτιά στην περίπτωση του Μάλι. Και αυτή είναι η ερώτησή μου. Δεν είναι ερώτημα για την ανθρώπινα δικαιώματα, το σεβασμό τους φιλοσοφικά και με τα φυσικά ερωτήματα. Όταν κάποιος είναι αντιμέτωπος με ένα τρομοκράτη πρέπει να υπάρχει κάποιος που να μπορεί να αντιμετωπίσει, όχι να του βάλουμε μπροστά του ένα νομικό κείμενο. Κύριε Ενάρτ, θα ήθελα να προσθέσω, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, αλλά φοβάμαι ότι η ερώτησή σας υπερβαίνει τον τομέα των καθηκόντων του κυρίου Μαριάννη. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, να θέσετε την ερώτηση αυτή στον αρμόδιο. Ή μπορούμε να τη θέσουμε στη διάρκεια κάποια συνεδρίασης με την κυρία Μογκερίνη για παράδειγμα. Σε μια συνάντηση εκεί. Και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω από τον κύριο Μπόρις Κορμανέτσι να λάβει το λόγο και μετά αν ο κύριος Μαριάννη θέλει να απαντήσει θα του δώσουμε και το λόγο μετά τον κύριο Κρυμινέτσκι. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Καταρχά, όσον αφορά την ποιότητα και την ποστή, όλε οι μονάδε που στέλνονται σε διεθνεί επιχειρήσει έχουν δύο στάδια πιστοποίηση. Εθνική πιστοποίηση και στη συνέχεια ε, για το ΝΑΤΟ. Ε, ή το ΝΑΤΟ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση για το ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε να δεχτούμε λοιπόν το επιχείρημα ότι δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένε οι μονάδε μα. Οι μονάδε που στέλνουμε είναι πλήρω επιχειρησιακέ και πλήρω κατάλληλε για αυτέ τι μορφέ επιχειρήσει. Δεύτερη ερώτηση για την υποστήριξη της Ουκρανίας με περισσότερα όπλα. Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Εμείς ε, συνεργαζόμαστε σε, διεθ... διμερές επίπεδο με τους συναδέλφους ε, σε θέματα στρατιωτικής και τεχνικής συνεργασίας, αλλά σας παρακαλώ μην λησμονείτε ότι η Ουκρανία είναι η μόνη χώρα στην οποία σκοτώθηκαν άνθρωποι ε, για ε, λόγους ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πέθαναν για τις ευρωπαϊκές αξίες και αυτό δεν θα πρέπει να το λησμονούμε. Δεύτερη ερώτηση. Πήρα από τις διεθνείς επιχειρήσεις. Σαφώς και χρησιμοποιούμε την πείρα μας καταρχάς ε, για την ε, αλλαγή και μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεών μας και αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο η εμπειρία, αλλά άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις ε, μονάδες μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σαφώς και συμμετέχουμε στην όλη έννοια των μονάδων μάχης, αλλά θα πρέπει κάτι να γίνει επιπλέον. Αυτή η έννοια των μονάδων μάχης θα πρέπει να χρησιμοποιεί για το σκοπό τον οποίο σχεδιάστηκε πριν από 10 χρόνια όταν δημιουργήθηκαν αυτές οι μονάδες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάννη, θέλετε να προσθέσετε κάτι στα όσα είπατε προηγουμένως. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εάν ε, δεν απάντησα η ερώτηση είναι πέραν ε, των ε, δικών μου των ορμοδιοτήτων, αλλά θα ήθελα τουλάχιστον να σας πω αυτά τα οποία έχω ακούσει ε, λόγω συμμετοχής μου σε συνεδριάσεις με τα Ηνωμένα Έθνη, διότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν και ρόλο αναφοράς ε, για την εκπαίδευση των μονάδων που εκπαιδεύονται στο Μάλι. Και το επίπεδο ικανοποίησής τους ήταν θετικό, έδωσαν θετικό βαθμό. Ε, όμως, πέραν αυτού, στο δεύτερο στάδιο της αποστολής UTM Mali υπάρχει ένα στάδιο επανεκπαίδευση όσο αποκαλείται. Λοιπόν, στρατεύματα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί, όταν επιστρέφουν περνούν μια δεύτερη διαδικασία εκπαίδευση και σε αυτή τη διαδικασία δεύτερης εκπαίδευση, οι ελλείψει και τα κενά τα οποία ε, έχουν επισημανθεί, διότι ε, να πούμε ότι η επιχείρηση ξεκίνησε μόλι πέρσι, Ξεκινούν μια δεύτερη εκπαίδευση λοιπόν, ε, όπου επικεντρώνονται σε τομείς στους οποίους υπήρξαν ελλείψεις. Αυτό είναι όλα όσα ξέρω να σας πω, αλλά σε περίπτωση που χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες, θα μπορούσα κάλλιστα να σας φέρω σε επαφή με τους αρμόδιους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε λοιπόν το σημείο αυτό και να ευχαριστήσουμε του ομιλητέ μας για την εξαιρετική εισαγωγή και απαντήσεις στη συνέχεια λοιπόν σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας είναι στις 5 Νοεμβρίου και με αυτό πέρασε τη συνεδρίαση.